Dear friends. Αγαπητοί φίλοι, θα ξεκινήσουμε παρακαλώ τη διάσκεψή μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσοι έχουν έρθει και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις ε, γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης Και πρέπει να βρείτε το σωστό κανάλι για να ακούσετε τη γλώσσα που μιλάτε, τη γλώσσα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική διάσκεψη με συμμετοχή των Ευρωβουλευτών και θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Ας, ε, Ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνο για την ισότητα των φίλων... χαίρομαι ιδιαίτερος που βλέπω τόσους πολλούς παρόντες εδώ, ενωμένους για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τείνουμε να θεωρούμε ότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα είναι ίσα, ισότιμα. Σε όλο τον κόσμο έχουν περισσότερες πιθανότητες ε, τα κορίτσια να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση από τα αγόρια και φαίνεται να έχουν και καλύτερες επιδόσεις στα πρώτα χρόνια του σχολείου. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δε πλειοψηφία τα κορίτσια πτυχιούχοι της ε, ανώτατης εκπαίδευσης. Συμφωνώ ωστόσο με την ε, Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τη Ισότητα των Φύλων ότι μπορεί να έχουμε αφήσει σε λανθάνουσα κατάσταση τη συζήτηση για τις αναπομένουσες ανισότητες ε, στην ε, εκπαίδευση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι διαφορετικές ακόμη οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες. Αλλά πιστεύω, όπως συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι πρέπει και καλά κάνουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές μεταξύ των ε, ε, εξαιρετικών επιδόσεων των κοριτσιών ε, μεταξύ αυτής της εξαίρετης επίδοσης ή ε, της παρουσίας των κοριτσιών στα σχολεία και των επιδόσεών τους στα μαθηματικά, τις επιστήμες ε, και τις επιλογές σταδιοδρομίας. Έχουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες από φύτους και στα μαθηματικά, τις επιστήμες, τεχνολογία. Τομείς δηλαδή που συνδέονται με τις καλύτερες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα λοιπόν και πρέπει να δούμε αν μπορούμε να το επιλύσουμε. Ίσως δεν μπορούμε να το επιλύσουμε άμεσα. Αισιόδοξος όμως παραμένω και ελπίζω ότι θα μπορέσει να λυθεί σύντομα. Επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε τις φωνές των ειδικών που έχουν έρθει εδώ να μας μιλήσουν, ώστε να δούμε πώς η κοινωνία συμπεριλαμβανομένων και των διδασκάλων επηρεάζει τις επιλογές ζωής των γυναικών, των κοριτσιών και γυναικών. Θέλω λοιπόν να ακούσω τις δικές τους εμπειρίες, εμπειρίες από τα κράτη-μέλη, τις εμπειρίες από τις χώρες της διεύρυνσης. Και ελπίζω, μετά τη συνεδρίασή μας, να αισθανθούμε όλοι ακόμη περισσότερο ισχυρή την προσήλωση για τη βελτίωση των ε, συνθήκων και την αντιμετώπιση των εναπομεινασών ε, προκλήσεων για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Περιμένω να ακούσω τα σχόλια και τα συμπεράσματα της διάσκεψης. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε κυρία Παπαδημούλη. Εκ μέρους ε, της Προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, που θα έρθει σε λίγο για να λάβει μέρος στη διάσκεψη, θα ήθελα να καλωσορίσω ε, τους συμμετέχοντες. Έχουμε 62 ευρωβουλευτές, άνδρες και γυναίκες, κυρίως γυναίκες βέβαια, από 18 χώρες μέλη και επιπλέον από την Ορβηγία και ε, από έξι χώρες ε, που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης. Πριν δώσω το λόγο στην Επίτροπο Γιώουροβα, που βρίσκεται εδώ και θα μας κάνει μια παρουσίαση, ε, έχω τη τιμή να σας παρουσιάσω ένα πολύ θαραλέο κορίτσι. Και ίσως είναι το καλύτερο παράδειγμα το κορίτσι αυτό και η πλέον κατάλληλη για να μας πείσει για τη σημασία που έχει ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση των κοριτσιών και των αγοριών. Γιατί έτσι, με τη μόρφωση θα χειραφετηθούν τα κορίτσια και οι γυναίκες. Ε, πέρυσι το κορίτσι αυτό βραβεύθηκε ως ε, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κορίτσι της Χρονιάς. Πιστεύω ότι έχει ένα σημαντικό μήνυμα να μας, ε, μεταφέρει Γι' αυτό δίνω το λόγο στη Μανών Βαν Χόρεμπεκ. Σας ευχαριστώ. Λέγομαι Μανών Βαν Χόρεμπεκ. Είμαι 11 ετών και τον Οκτώβριο βραβεύτηκα με το βραβείο ψηφιακό κορίτσι της χρονιάς γιατί ασχολούμαι με την τεχνολογία και θέλω να έχουν όλο και περισσότερα κορίτσια πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Φέτος ε, ξεκίνησα το γυμνάσιο και ήταν για μένα ένα μεγάλο βήμα αυτή η μετάβαση. Γιατί πέρασα από ένα σχολείο που είχαμε smartboards και υπολογιστές σε κάθε μάθημα και ήταν μεγάλο βήμα αυτή η μετάβαση στο γυμνάσιο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μήνυμα λοιπόν που θα ήθελα να σας διαβιβάσω εδώ σήμερα είναι ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι το μέλλον και οι τεχνολογίες το ίδιο. Τεχνολογίες βρίσκουμε παντού, στα έξυπνα τηλέφωνα, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητα. Είναι σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της ζωής μας. Και μάλιστα είναι σημαντικό στα γυμνάσια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να έχουμε περισσότερα μαθήματα για τις νέες τεχνολογίες για να μπορέσουμε με ευρηματικό και δημιουργικό τρόπο να βρούμε λύσεις ε, και να βρούμε τα κλειδιά για τα προβλήματά μας. Είναι σημαντική λοιπόν η τεχνολογία στα σχολεία. Και μάλιστα ε, είναι εδώ μια φωτογραφία από την πρώτη μέρα που παρακολούθησα μάθημα προγραμματισμού. Ήταν πραγματικά καταπληκτική ε, εμπειρία, ενθουσιάστηκα και λέω μπορώ κι εγώ να κάνω προγραμματισμό. Γιατί έτσι θα μπορέσω να προγραμματίσω και να κατασκευάσω ακόμη και μικρά ρομπότ συναρπαστική εμπειρία. Και εδώ βλέπετε στη φωτογραφία αυτό που κατασκεύασα, το πρώτο μου ρομπότ. Το πρώτο μου ρομπότ ε, το κατασκεύασα στην ηλικία των 8 ετών. Ήταν η πρώτη μου επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Τώρα είμαι και προπονήτρια, εκπαιδεύτρια για παιδιά. Ε, μαθαίνω προγραμματισμό και κωδικοποίηση στα άλλα παιδιά και τα βοηθάω όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα Και στη φωτογραφία αυτή εκπαιδεύσαμε εργαζόμενους σε μια μεγάλη επιχείρηση στο θέμα του προγραμματισμού. Γιατί δεν ήξεραν τις δυνατότητες που δίνει ο προγραμματισμός και μέσα σε μία μέρα οι εργαζόμενοι αυτοί κατάφεραν να μάθουν τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού. Εδώ είχαμε μία συνάντηση με την Έλλη Κρούς. Η Έλλη Κρούς είχε την ιδέα να κάνει μερικές πεταλούδες να πετάξουν τεχνητές. Είχε την ιδέα, αλλά δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να το καταφέρει κιόλα. Και μετά από μία μέρα και πολλές προσπάθειες κατάφερε να υλοποιήσει αυτή τη την ιδέα. Παρόλο που ήταν απεσιόδοξη στην αρχή. Μέσα σε μια μέρα τα κατάφερε. Και ήταν ενθουσιασμένη με αυτή τη την επιτυχία. Επίσης θα ήθελα να απευθύνω και μία έκκληση σε εσά τους ευρωβουλευτές γιατί πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι πραγματικά απαραίτητη και χρειαζόμαστε μαθήματα τεχνολογίας ήδη από το γυμνάσιο. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας μιλήσω και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Έχω και blog στο ίντερνετ Ευχαριστώ, Μανών. Φαντάζομαι θα έχει λαμπρό μέλλον. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, αρμόδια Επίτροπο για την Δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων. Ε, ο λόγος στην Επίτροπο Βέρα Γιαούροβα. Αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, Αγαπητοί εθνικοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, πριν να αρχίσω και να λέω αυτό που ήθελα να πω σήμερα, θα ήθελα να εκφράσω τη ε, χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ και επίσης όταν άκουγα την Μανών έπρεπε να παραδεχτώ ότι ε, ε, εγώ ίδια δεν μπορούσα να θυμηθώ πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που είδα τελευταία φορά ένα παιδί περιτριγυρίζουμε από σοβαρούς ενήλικες όλη την ώρα. Πολύ καλό για ένα πολιτικό να περιτριγυρίζεται μόνο από σοβαρούς ενήλικες. Επειδή και εγώ είμαι μια σοβαρή και ενήλικη γυναίκα, οπότε είναι καλή αυτή η στιγμή όταν ακούμε, ερχόμαστε σε επαφή με τη νέα γενιά, τους νέους, τα νεαρά κορίτσια που αντιμετωπίζουν, αναλαμβάνουν τέτοιες προκλήσεις και Ελπίζω ότι κάποια κορίτσια βλέπουν τον εαυτό τους στον κόσμο της τεχνολογίας, γιατί ο κόσμος της τεχνολογίας πιθανότατα θα είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις, ε, τις συνθήκες διαβίωσης ε, στην Ευρώπη και θα χρειαστούμε τέτοια νεαρά κορίτσια. Σας ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό κυρίες και κύριοι τώρα για την παραμονή της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας. Ε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι μαζί σας για να γιορτάσουμε τα ε, επιτέγματα μας όσον αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχουμε σημειώσει εξωσημείωτη πρόοδο προς τη συνισότητα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Έχουμε συνδυάσει τους πόρους μας και τα μέσα μας νομικά, πολιτικά και οικονομικά ώστε να επιφέρουμε αλλαγές. Η νομική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό και αυτό μάλιστα χάρη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σε μεγάλο βαθμό. Οι, γυναίκες δεν μπορούν να υπόκειται σε διακρίσεις επί τη βάση φύλου, ε, κοινωνικής ασφάλισης και πρόσβασης ε, στα ε, αγαθά και τις υπηρεσίες. Ε, ε, αυτή είναι η νομοθεσία, τώρα δικό μας έργο είναι να την υλοποιήσουμε. Στην Ευρώπη ε, θα τις γυναίκες να εργάζονται. Ε, αυτό είναι ο ρόλος της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής ανεξαρτησίας. Ε, έχουμε εργαστεί ώστε να υπάρχει ισορροπία εργασιακής ζωής για τις γυναίκες και για τους άνδρες. Γι' αυτό και έχουμε φτιάξει νομοθεσία για τη γονική άδεια, για τη μερίμνα των παιδιών, αλλά και για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια από την βία που οφείλεται στο, στη διαφορά φύλου. Επίσης στηρίζουμε τις εθνικές κυβερνητικές εκστρατείες καθώς και τα προγράμματα κατά της βίας με βάση το φύλο. Σήμερα οι γυναίκες είναι πολύ μορφωμένες, πολύ περισσότερες γυναίκες εργάζονται από ό,τι παλιότερα. Ε, Είμαστε καινοτόμες ε, και ε, έχουμε επιχειρηματικό πνεύμα. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ε, να προχωρήσουν σε σταδιοδρομίες, στις επιστήμες και στην τεχνολογία της ενημέρωσης. Ακούσαμε μόλις την Μανώνα, το την... Το την Ευρωπαία ψηφιακή κοπέλα, ε, συγχαρητήρια και πάλι. Ε, θέλουμε να σας, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα όμως για τις προκλήσεις που παραμένουν μπροστά μας. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα PISA, η Οι διαφορές του φίλου στην, στα μαθηματικά αλλά και σε, ε, σε, άλλα μαθήματα ε, μειώνονται. Ωστόσο, όταν τα παιδιά είναι γύρω στα 15, τα κορίτσια φαίνεται να είναι πιο αγχωμένα για τα μαθηματικά και λιγότερο, να έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση. Ε, ωστόσο, οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται λιγότερο στη μηχανική, στις επιστήμες και στα μαθηματικά, ενώ οι άνδρες είναι περισσότεροι απόφοιτοι, ε, σε τελειόφοιτοι σε αυτούς τους τομείς. 60% στους μηχανικούς, ε, στις επιστήμες και στα μαθηματικά είναι άνδρες. Ακόμα και αν οι γυναίκες αποφοιτούν σε αυτές τις, θετικέ θετικές επιστήμες, λιγότερο πιθανό είναι να εργαστούν σε αυτούς τους τομείς. Δύο φορές είναι οι άντρες περισσότεροι από τις γυναίκες που εργάζονται στην έρευνα και στην ανάπτυξη. 2,6 εκατομμύρια άνδρες σε αντίθεση με 1,3 εκατομμύρια γυναίκες που αντιπροσωπεύουν κάτω από το 20% στους, ε, των μηχανικών και των μηχανικών υπολογιστών. Είναι ατυχές που χάνουμε τέτοια ταλέντα στις επιστήμες που χρειαζόμαστε στην αγορά εργασίας και μόνο με τις γυναίκες και το δικό τους ταλέντο θα μπορέσει η Ευρώπη να είναι οικονομικά ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έχουν ρόλο κλειδί να παίξουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων τα βιβλία τα, θα πρέπει να ε, αντιπαρέρχονται, να αντιπαρατίθενται στα στερεότυπα του τύπου και με τον συνάδελφο Ναύρατζη θέλουμε να δουλέψουμε ώστε να προωθήσουν τα σχολεία την ισότητα των φύλων. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Τα περισσότερα κορίτσια και τα αγόρια έχουν συμπεριφορές, προσδοκίες και όνειρα ε, θέλουν να ενταχθούν στην κοινωνία και στην οικονομία, ωστόσο βλέπουν ότι υπάρχει ανισότητα και κάποιες φορές και βία. Και άρα τα μαθήματα για την, ε, τον σεβασμό και την ισότητα δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Ένας δάσκαλος μπορεί να λέει στη γόρη σας να είναι φιλόδοξη και αισιόδοξη, όμως αργότερα 60% λιγότερο θα πληρώνετε από ότι οι άντρες ε, συμμαθητές της. 16 λιγότερο θα πληρώνεται από ότι οι άντρε μαθητέ τη. Ενώ μπορεί να αποδίδει και περισσότερο από εκείνου. Και πιθανότατα θα εργαστεί σε μερική απασχόληση, θα διακόψει τη σταδιοδρομία τη για να φροντίσει άλλους. Και δεν θα έχει πολλέ πιθανότητες να ανέβει στην κλίμακα την ε, εργασιακή, θα μείνει στο 40% χαμηλότερα από ότι τα αγόρια συμμαθητέ τη η κόρη σας μπορεί κάποια μέρα να πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην εργασία ή στα παιδιά, ενώ ο σύζυγός σας θα μπορεί να πάρει γονική άδεια απλά για λίγο διάστημα. Αυτά είναι προβλήματα και διλήμματα και πρέπει να, ε, να, επιτείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε οι κοινωνικοί εταίροι, οι τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις, τα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα εκπαιδευτικά και ε, ε, ιδρύματα να εργαστούν υπέρ της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη. Εγώ θέλω να στηριχτούν οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των κρατών μελών και όλοι οι οι φορείς να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους ε, για την απασχόληση την ε, σύνταξη και τη λήψη αποφάσεων και περισσότερες γυναίκες σε αυτούς τους τομείς. Ε, πρέπει επίση να επιταθούν οι προσπάθειες ώστε να καταπολεμηθεί η βία με βάση το φύλλο. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικιακής βίας είναι ένα καλό σημείο κίνησης για όλους μας και τα κρατημέλη μας θα πρέπει να την επικυρώσουν. Εγώ θα εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αποτελεί μια καλή ε, διεύθυνση για τις Ευρώπες και θα λάμπει ως πρότυπο παγκοσμίω για την υπεράσπιση των ε, ίσων δικαιωμάτων. Θα στηρίξουμε τη χειραφέτηση των γυναικών και των ε, κοριτσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις χώρες που είναι υποψήφιες για την προσχώρηση στην Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Γυναικών ιδιαίτερα για την ε, προσήλωσή σας στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Και είμαι ευτυχής που εορτάζουμε τη, μαζί την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας σήμερα και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιώργοβα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την συνέντευξη τύπου, κοινή συνέντευξη τύπου 12 και 30. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους ε, και τις βουλευτές που βρίσκονται στο, στην ε, αίθουσα. Θα παρακολουθήσουμε τώρα μία, ένα μήνυμα μαγνητοσκοπημένο της ε, δόκτωρος Χαουά Ιμπραχήμ. Ξέρετε ότι υπογραμμίζει την σημασία της εκπαίδευσης στη χειραφέτηση των γυναικών. Άλλο ένα ορόσημο, άλλος ένας χρόνος. Χαιρετίζουμε το 50% γυναίκες αυτή την ε, Διεθνή ημέρα των γυναικών 2015. Το θέμα του Ευρωπαϊκού, που επέκρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η χειραφέτηση των γυναικών ε, και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης καταλληλότερη στιγμή δεν μπορούσε να διαλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια. Εγώ γεννήθηκα στο βορειοανατολικό κρατήδιο, κράτος της Νιγηρίας, σε ένα χωριό που ονομάζεται Χίναχ, ε, τυχαία πήγα σχολείο, τυχαία έγινα δικηγόρος, τυχαία επελέγει να διδάξω στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ. Τώρα βρίσκομαι στο χασιμητικό βασίλειο της Ιορδανίας, κατόπιν προσκλήσεως ε, του ε, η του πρίγκιπα Χασάν ε, και πιστεύω ότι και αυτό τυχαίο είναι. Αλλά αυτή η τύχη που μου προσέφερε ζωή δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εκπαίδευση, χωρίς την παιδεία. Αυτό που χαιρετίζουμε σήμερα λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε εκατομμύρια κορίτσια που δεν είχαν ε, την ευκαιρία να πάνε στο σχολείο αυτή την ευκαιρία πρέπει να τους προσφέρουμε. Ας διαρωτηθούμε, λοιπόν με τη ειλικρίνεια, ας θέσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του ερωτήματος τι άλλο μπορώ να κάνω, τι άλλο μπορώ να δώσω για να εξασφαλίσω σε ένα ακόμα παιδί την εκπαίδευση. Έχουμε κάνει πολλά και συνεχίζουμε. Επιπλέον όμως τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να βάλουμε στο πρόγραμμά μας, στο στόχο μας, μια εκπαίδευση ανοιχτή σε όλα τα παιδιά, μια εκπαίδευση που θα περιλαμβάνει και τη θρησκεία και την παράδοση και που θα στρέφεται προς τις νέες τεχνολογίες και προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια ολιστική εκπαίδευση των κοριτσιών. Σκέφτομαι έναν κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας τώρα, τον κίνδυνο της τρομοκρατίας και τον κίνδυνο των εξτρεμισμών. Τα κορίτσια αυτά είναι εκείνα τα οποία θα προσδιορίσουν το μέλλον μας. Και πιστεύω ότι αν επενδύσουμε στα κορίτσια αυτά, επενδύουμε στην ε, ανθρωπιά μας που ακόμα δεν έχει γεννηθεί. Και στην ανθρωπότητα που δεν έχει γεννηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να πω για άλλη μια φορά ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σε απευθύνω τον λόγο. Σας εύχομαι πολύ επιτυχημένες εργασίες στη Διεθνή ημέρα της γυναίκας 2015. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας λοιπόν για να... και, και ας χαιρετήσουμε, ας επιδείξουμε αυτήν την αντοχή στους αγώνες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη μεταβίβαση των αξιών της αγάπης και της συγχώρησης για τις γενιές που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί. Bueno, pues para final... Ωραία. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο γύρο παρουσιάσεων, θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά την ε, Επίτροπο την κυρία Γιώροβα και τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη, και να τους απελευθερώσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν το κοινοβουλευτικό τους έργο και τις κοινοβουλευτικές τους υποχρεώσεις. Τους ευχαριστώ θερμά που είχαν την καλοσύνη να έρθουν στην, κατά την έναρξη της διάσκεψης αυτής και εμείς να περάσουμε στο πρώτο πάνελ, στην πρώτη θεματική ενότητα αυτής της διάσκεψης. Και όσο περιμένω τους καλεσμένους μας στο πρώτο πάνελ να ανέβουν στο Προεδρείο, να σας ενημερώσω για μερικά διαδικαστικά για να μπορέσετε να ζητήσετε το λόγο και να μιλήσετε μετά την παρουσίαση των καλεσμένων μας, πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο. Για τους ευρωβουλευτές ε, ισχύει η κανονική διαδικασία, η συνηθισμένη. Μπορούν να ζητήσουν το λόγο. Οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο που έχουν μπροστά τους με διαφορετικά χρώματα. Βλέπετε τους κλητήρες στους διαδρόμους θα συγκεντρώσουν τα έντυπα που έχετε συμπληρώσει ότι ζητάτε το λόγο. Έχουμε χρησιμοποιήσει διαφορετικά χρώματα για να ξέρουμε για ποιο πάνελ ζητάει το λόγο ο κάθε προσκεκλημένος. Για την πρώτη συζήτηση θα συμπληρώσετε το γαλάζιο έντυπο, για τη δεύτερη το ροζ και για την τρίτη το κίτρινο. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε να λάβετε το λόγο στην πρώτη θεματική ενότητα, συμπληρώστε το γαλάζιο έγγραφο. Αν θέλετε το λόγο στη δεύτερη θεματική ενότητα, το ροζ έγγραφο. Και στην τρίτη, το κίτρινο έγγραφο. Οι παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία λεπτά. Για να δώσουμε το λόγο σε όσο το δυνατό περισσότερους ομιλητές. Αυτά ως προς τα διαδικαστικά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να ζητήσετε και να λάβετε το λόγο. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη μας θεματική ενότητα και να δώσω το λόγο στον κύριο Κόρη, που είναι ο Διευθυντής ε, του Γραφείου της UNICEF στις Βρυξέλλες και θα μας παρουσιάσει το χάρτη των δικαιωμάτων των παιδιών. Κύριε Κόρη, σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε την καλοσύνη να έρθετε στην συνεδρίασή μας, στη διάσκεψη αυτή για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί Μανών, αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής τη Ισότητα των Φύλων και των Δικαιωμάτων τη Γυναίκα, τη κυρία Καρσία Πέρε, και τη Προέδρου τη ε, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία, τη Σίλβια Κώστα, για το ότι τόνισαν τη σημασία που έχει η χειραφέτηση των κοριτσιών μέσω τη μόρφωση. Έτσι, ε, σηματοδοτούμε αυτή τη Διεθνή μέρα της γυναίκας. Για κάθε παιδί, κάθε κορίτσι, παντού, η, η μόρφωση δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα, είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα και η πρόσβαση στο δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να περιορίζεται ούτε από σύνορα, ούτε από εισόδημα, ούτε καν από, μια, από κάποια αναπηρία. Ούτε θα πρέπει το μέλλον του παιδιού να περιορίζεται από το φίλο του, επειδή είναι κορίτσι δηλαδή. Σε χαλεπούς οικονομικούς καιρούς ε, πολύ συχνά το κορίτσι θα είναι το πρώτο που θα εγκαταλείψει το σχολείο, πολύ νωρίτερα από τα αδέρφια του. Αν και όλα μπορέσει να πάει σχολείο. Μπορεί να περιμένει ένα κορίτσι ε, πολύ χαμηλότερες αποδοχές από τους άνδρες ε, συναδέλφους της. Αν υποθέσουμε ότι θα έχει δικαίωμα σε οποιοδήποτε μισθό χωρίς ε, μια ποιοτική στοιχειώδη μόρφωση, κατά πάσα πιθανότητα το κορίτσι θα παντρευτεί πολύ νωρίς και μάλιστα παρά τη βουλησή της, πολύ πιθανό να, να πεθάνει κατά τη διάρκεια του τοκετού και μάλλον απίθανο να, έχει, να αποκτήσει υγιή παιδιά και να μπορέσει να τα στείλει στο σχολείο. Έτσι διαιωνίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος ε, της διακριτικής μεταχείρισης. Υπάρχουν συντριπτικά και αδιάστητα στοιχεία ότι η πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει τα ίδια τα κορίτσια αλλά και τις κοινότητες, τις κοινωνίες ε, που, στις οποίες ζουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, κορίτσια με πολλά χρόνια μόρφωσης ε, παντρεύονται τέσσερα χρόνια αργότερα και έχουν λιγότερα παιδιά, κατά 2,2 λιγότερα παιδιά. Και μάλιστα μία μελέτη σε 50 χώρες δείχνει ότι κάθε επιπλέον χρονιά φοιτησης σε μία χώρα αυξάνει το ΑΕΠ, το, το ΑΕΠ 40 ετίας της χώρας κατά 0,37 μονάδες. Και μάλιστα μια μορφωμένη μητέρα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να στείλει και τα παιδιά της στο σχολείο. Η χειραφέτηση λοιπόν των κορισιών μέσω τη μόρφωσης θα προκαλέσει μεγάλες αλλαγέ και σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο γενιάς. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν πολλά εμπόδια και πολλοί φραγμοί που παρεμποδίσουν την πρόοδο, με παλιές και νέες προκλήσεις για τα κορίτσια παντού, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Πώς μια οικογένεια θα στείλει το κορίτσι της στο σχολείο με τόσο υψηλό κόστος εκπαίδευσης. Και τι γίνεται με τα στερεότυπα για το γυναικείο ρόλο ακόμη και με μόρφωση. Πώς μπορούν τα κορίτσια να αποκτήσουν την πρακτική εμπειρία που χρειάζονται για να βρουν δουλειά. Πώς ε, θα εξασφαλίσουμε να ενημερωθούν τα κορίτσια για τα δικαιώματά τους. Γιατί αυτά τα ζητήματα αφορούν τα κορίτσια παντού και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η UNICEF συνεργάζεται με αναπτυσσόμενες χώρες και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αναζητώντας ε, καινοτόμους ε, και εύχρησους τρόπους για να ανταποκριθεί στις ε, προκλήσεις ε, ως προς τα δικαιώματα των κορίσιων και την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνοντας γνώση, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση στα κορίτσια για να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τους, όπως μας απέδειξε πριν από λίγο η Μανών, να βελτιώσουν την ε, πολιτική και κοινωνική τους συμμετοχή και να πιστέψουν στις ικανότητές τους, είναι ένας στόχος ε, που θα υλοποιηθεί μόνο αν προωθήσουμε ε, με δυναμικό και δραστήριο τρόπο τα δικαιώματα των παιδιών και των κοριτσιών. Μάλιστα έχουμε δημιουργήσει μια ε, εργαλειοθήκη για τα δικαιώματα των παιδιών βάζοντας στο επίκεντρο όλα τα παιδιά και τα κορίτσια, στο επίκεντρο των μαθησιακών προσπαθειών. Έτσι θέλουμε να χειραφετήσουμε όλα τα παιδιά και τα κορίτσια μέσω της μόρφωσης. Μάλιστα σας έχουμε μοιράσει και ένα φυλάδιο για την εργαλειοθήκη αυτή με πληροφορίες ε, για το πρόγραμμα αυτό της UNICEF. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω εδώ την, ε, τον παραλληλισμό με ένα δέντρο όταν μιλώ για την εργαλειοθήκη. Πρόκειται για ένα δέντρο με τρία κλαδιά. Τα κορίτσια θα πρέπει να μπορέσουν να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους, το ένα κλαδί, μέσω των δικαιωμάτων τους, ε, το δεύτερο κλαδί και με σκοπό να αποκτήσουν δικαιώματα. Είναι το τρίτο κλαδί. Εκατοντάδες σχολεία στην Ευρώπη χρησιμοποιούν αυτή την καινοτόμα προσέγγιση χαμηλού κόστους με εντυπωσιακά αποτελέσματα, ακόμη και σε απρόσφορο έδαφος μερικές φορές. Η πρόθεση της ένταξης των κορισιών σε προγράμματα ε, σπουδών, σε σχολικά βιβλία και σε μαθησιακό υλικό είναι βασική και μεθοδολογία για την υλοποίηση της ισότητας των δύο φύλων. Και αυτό είναι το πρώτο κλαδί του δέντρου για τα δικαιώματα των παιδιών. Η μάθηση για τα δικαιώματα. Και μάλιστα αυτό θα ήθελα να συμπεριληφθεί και στο, στην έκθεση που ετοιμάζει ο Δ. Ροντρίγκε στην Επιτροπή Γυναικών. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα η μάθηση μέσω των δικαιωμάτων σημαίνει τροποποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος ώστε τα δικαιώματα αυτά να τα βιώνουν καθημερινά, ως καθημερινή εμπειρία τα παιδιά και να μην περιορίζονται μόνο στο αντικείμενο ενό μαθήματο. Για παράδειγμα, ο σεβασμό των δικαιωμάτων των κοριτσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στι πολιτικέ των σχολείων και σε μηχανισμού για την προώθηση τη δημοκρατική συμμετοχή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για να υλοποιήσουμε την ισότητα των φύλων στα σχολικά συμβούλια θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα στα σχολικά συμβούλια και κορίτσια και αγόρια. Επίσης, ε, η μάθηση μέσω των δικαιωμάτων να μας οδηγεί στη μάθηση με σκοπό τα δικαιώματα. Δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά να εντοπίζουν ε, δικαιώματα που τους ενδιαφέρουν. Είδαμε το παράδειγμα της Μανών. Και επίσης δραστήρια να προσπαθούν για την υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων σε τοπικό, σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι τα σχολεία θα πρέπει να δημιουργήσουν πρόσφορες συνθήκες για κριτική σκέψη, προθώντας ε, την ισότητα των φύλων και ε, καλλιεργώντας και τροφοδοτώντας σχετική συζήτηση. Και στο σημείο αυτό, περισσότεροι θέσμες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη ε, θα μπορούσαν να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η χειραφέτηση των μέσω της Μορφωση είναι σημαντική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσουμε από την συγκέντρωση που έχουμε στην ποσότητα, στη συγκέντρωσή μας στην ποιότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 83% των νεαρών κοριτσιών φτάνουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών 78%. Επίσης 60% των αποφύτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες. Βέβαια, μερικές φορές η ποσότητα επισκιάζει τους βασικούς στόχους της υλοποίησης ε, της ισότητας των δύο φύλων, που είναι η ποιότητα. Γι' αυτό και θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα σχολεία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Και τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις πτυχές ε, της διαπαιδαγώγησης που δίνεται μέσα στο σχολείο και να μην περιορίζονται σε ένα πρόγραμμα ή σε ένα μάθημα. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο 3.300 σχολεία αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί στο βραβείο των σχολείων που σέβονται τα δικαιώματα. Και αυτή η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα υποφελής και για τα παιδιά, ιδιαίτερα τα κορίτσια, αλλά και για τους δασκάλους, τους γονείς, τις οικογένειες και γενικότερα, γενικότερα την κοινωνία. Οπότε θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις παλιές μαθησιακές μεθόδους και να βελτιώσουμε τα σχολεία, να έχουμε σχολεία που δεν θα αποκλείουν να βελτιώσουμε τις μαθησιακές τεχνικές, τα προγράμματα σπουδών και να καταπολεμήσουμε τα χάσματα και τις διαφορές ε, καθώς και τα στερεότυπα. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις ε, στην πρόορη και την προσχολική ε, εκπαίδευση και αν θέλουμε μια κοινωνία με ισότητα των δύο φύλων, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Και αν θέλουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που έχει χειραφέτηση των γυναικών, θα πρέπει να δουλέψουμε ταυτόχρονα όχι με κορίτσια και γυναίκες μόνο, αλλά και με αγόρια και άντρες, με ηγέτες, πολιτικούς, ηθήνοντες, με φορείς, σχολεία και όσους έχουν επίδραση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική σφαίρα. Η χειραφέτηση, το empowerment, ακούγεται πολύ τον τελευταίο καιρό. Όταν λέμε empowerment, αυτή η χειραφέτηση εμπεριέχει και τον όρο power, την εξουσία, που είναι μια, ένα πολύ σημαντικό αγαθό ε, και ακούγεται πάρα πολύ και όταν μιλούμε για empowerment στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, το να δώσουμε εξουσία στις γυναίκες, πιστεύουμε ότι πραγματικά αυτή η ισορροπημένη κατανομή της εξουσίας είναι το σημαντικότερο φάρμακο για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες. Βέβαια, η εξουσία μερικές φορές είναι απρόσιτη για πολλά κορίτσια και γυναίκες, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα κορίτσια και για τα παιδιά παντού, τι σημαίνει εξουσία. Εξουσία σημαίνει να μπορεί κανείς να λαμβάνει ελεύθερα τις αποφάσεις του και τεκμηριωμένα να είναι ισότιμος εταίρος, να μπορεί να συμμετέχει στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο νοικοκυριό του, στο σπίτι του, αλλά και στην κοινωνία όταν έλαβε το βραβείο Ζαχάροφ το 2013, η Μαλάλα Ιουσουφζάη μας εξήγησε πολύ εύγλωτα και γλαφυρά γιατί είναι σημαντικός ο αγώνας της για την μόρφωση. Θα παραθέσω αυτά που είπε στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια. Μία χώρα θα πρέπει να κρίνεται ως προς την ισχύ της, όχι από τον αριθμό των ε, στρατιωτών της και του ναυτικού της. Θα πρέπει η ισχύ της να κρίνεται με βάση τα ποσοστά αλφαβητισμού. Θα πρέπει να κρίνεται με τον αριθμό των μορφωμένων ανθρώπων και από το κατά πόσο χορηγεί ε, βασική πρόσβαση στην ε, παιδεία, ισότητα μεταξύ των ανδρών και γυναικών γιατί πραγματικά μια χώρα με ταλαντούχους επιδέξους και μορφωμένους ανθρώπους είναι μια πραγματική υπερδύναμη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στα παιδιά, να επενδύσουμε στη μόρφωση, στην παιδεία και να εθετήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα σχολεία στην, ε, στα δικαιώματα των παιδιών προς την παιδεία. Και αυτό είναι μια ευκαιρία που δεν έχουμε την πολιτεία να χάσουμε. Όπως είπε και η Χάουα Ιμπραχήμ, δεν θα πρέπει η πρόσβαση στην ε, μόρφωση να γίνεται κατά τύχη. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. for your work. Σας ευχαριστώ κύριε Κόρη για τα λόγια σας. Είναι νομίζω σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι η παιδεία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γιατί ακριβώς μπορεί να αλλάξει και το μυαλό. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Ε, ομιλητρία. Την Ιβ Ένσλερ, που είναι Αμερικανίδα συγγραφέας και ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας που είναι γνωστή για το θεατρικό της έργο «Δύο μονόλογοι» και ενό παγκόσμιου κινήματο ε, για την ε, πάυση τη βία κατά των γυναικών. Καλημέρα σε όλου. Είμαι πολύ ευτυχή που βρίσκομαι σήμερα εδώ και μιλώ για την χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω τη ε, καλλιέργεια και τη παιδεία του. Ακούστηκαν ήδη πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα το πρωί Κάτι το οποίο πολύ σκέφτομαι τελευταία είναι όλα τα χρόνια που δούλεψα για να σταματήσω τη βία κατά των γυναικών. Έχουν περάσει 20 χρόνια, έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο, 70 χώρες περίπου και τελικά κατέληξα στο ότι όντως η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την βία. Και ταυτόχρονα όμως η βία επηρεάζει την εκπαίδευση των κοριτσιών. Πιστεύω ότι η παιδεία είναι το ξύφος που κόβει την ανισότητα. Το, το σπαθί που μπορεί να κόψει την, ε, περικόψει την ε, ανισότητα. Αλλά το κλειδί είναι η εκπαίδευση των κοριτσιών, γιατί όχι μόνο είναι παθιασμένα και έξυπνα τα κορίτσια, αλλά είναι και πολύ γενναιόδερα. Και όταν μαθαίνουν, ε, διαχέουν τη γνώση τους σε όλη τους την κοινότητα. Όταν εκπαιδεύεις λοιπόν ένα κορίτσι, εκπαιδεύεις και όλη τη την κοινότητα, την μικρή της κοινωνία. Να μιλήσω όμως και για τη βία, όπου και στην Ευρώπη ισχύει, όπου υπάρχει εκφοβισμός, παρενόχληση, σεξουαλική ε, ε, παρενόχληση ε, ε, ε, ακόμα και ακροτηριασμός γενετικών οργάνων και στη ΣΥΠΑ το ίδιο 300.000 κορίτσια, κορίτσια δέχονται επιθέσεις στα πανεπιστημιακά κάμπους στην Αμερική. Ε, βλέπουμε ότι βασικά αυτό που χρειάζονται λοιπόν οι γυναίκες είναι η ε, παιδεία. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις διασυνδέσεις ανάμεσα στην παιδεία και στη βία κατά το γυναικών. Να σας πω αυτό που πιστεύω βαθύτατα. Όπως είπα, έχω ταξιδέψει πολλά πολλά χρόνια σε πολλές χώρες και έχω δει ποιος είναι ο πυρήνας της βίας. Και για να είμαι ειλικρινή, πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για την έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγηση. Είναι δύσκολο να το συζητήσει αυτό κανείς οπουδήποτε στον κόσμο, ακόμα και εδώ στην Ευρώπη. Αν όμω δεν μάθουμε στα παιδιά και στα, στα αγόρια και στα κορίτσια τι είναι υγιεί σεξουαλικές σχέσεις, τι, τι σημαίνει συνένεση, τι σημαίνει βεβαιότητα ε, ε, σε πολύ πολύ μικρή ηλικία δεν τους μαθαίνουμε την ισότητα. Γιατί πάρα πολλά από τα όσα συμβαίνουν στις γυναίκες, στα κορίτσια, στη διάρκεια της παιδείας τους, της εκπαίδευσής τους, είτε έχουν να αντιμετωπίσουν επιθετικό εκφοβισμό ή σεξουαλική παρενόχληση, αν δεν έχουν μάθει τι θα πει ε, σεξ σε, χαμηλό, σε μικρή ηλικία δεν θα μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τη. Στο Κονγκό, θα σα πω ένα παράδειγμα, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα που λέγεται «Η πόλη της χαράς» ε, με μια καταπληκτική γυναίκα συνεργάτη δαϊκή. Έχουν έρθει εκεί γυναίκες που έχουν επιβιώσει από ακραία βία που οφείλεται στο φύλλο. έχει το πρόγραμμα αυτό και ένα τεράστιο συστατικό σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης όπου τα κορίτσια μαθαίνουν ε, το σώμα τους, ε, πια αρχίζουν να, μαθαίνουν, να κοιτούν τον εαυτό τους, να σέβονται το σώμα τους, ε, ε, και δεν μπορώ να σας πω πόσο ριζικά έχει επηρεάσει το πρόγραμμα αυτό κάθε πτυχή της παιδείας τους. Γιατί πολλά κορίτσια που έρχονται εκεί σε αυτό το πρόγραμμα δεν γνωρίζουν καν ότι είναι οι κύριες του σώματός τους, του σώματός τους, ότι έχουν το δικαίωμα να πούν όχι. Δεν ξέρουν καν πώς είναι φτιαγμένο το σώμα τους. Και αυτή η, η μόρφωση επηρεάζει όλη την υπόλοιπη μόρφωσή τους σε αυτή την πόλη της ε, χαράς. Ε, συνάντησα μάλιστα ένα κορίτσι ένα χρόνο μετά ε, και τους, ζήτησα, τους ρώτησα μετά από ένα χρόνο ποιες, πώς ήταν οι σχέσεις τους και είπαν όχι. Μάθαμε στην πόλη της Χαράς ότι πρέπει να εκτιμούμε τον εαυτό μας και να σκεφτόμαστε την μόρφωσή μας, την ανεξάρτησή μας και όταν βρίσκουμε αγόρια που είναι ίσα μαζί μας και που μας εκτιμούν, τότε θα ξεκινήσουμε μια σχέση. Και δεν τους βρήκαμε ακόμα. Και εγώ πίστεψα ότι ήταν, ε, θεώρησα ότι ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό, γιατί ε, εφόσον συζητήσαμε τη σεξουαλικότητα, μάθαν τα δικαιώματά τους και δεν μπορούμε να χωρίσουμε, να διακρίνουμε την παιδεία των αγοριών και των κοριτσιών από αυτό, από το να μάθουν δηλαδή τα δικαιώματά τους, την σεξουαλικότητά τους. Νομίζω ότι ε, φοβόμαστε να μιλήσουμε για το σεξ, αλλά πάρα πολλά σημαντικά πράγματα που οδηγούν στη βία οφείλονται στην ε, μη κατανόηση του σεξ. Τα αγόρια δεν ξέρουν τι είναι το σεξ, επιτίθενται στα κορίτσια, επιδάν πάνω τους ξαφνικά, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν τι θα πει. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν την ντροπή και να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Τελειώνοντας να σας πω ότι πιστεύω ότι μιλάμε για πολύ για την εκπαίδευση των κοριτσιών, αλλά κάτι το οποίο δεν σκεφτόμαστε είναι οι μακροπρόθεσμοι ε, σε επιπτώσεις του να μην εκπαιδεύονται τα κορίτσια. Ε, εάν δεν μάθουμε στα κορίτσια αρκετά νωρί ότι έχουν το δικαίωμα να μάθουν, <clears throat> να είναι, ότι έχουν το δικαίωμα να γίνουν επιστήμονες, ηγέτες, ότι πρέπει να μάθουν να είναι κυρίες του εαυτού τους, αλλά και ταυτόχρονα έχουν το δικαίωμα να είναι και μητέρες, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και όταν είναι μορφωμένα τα κορίτσια, πολύ συχνά ε, παρατούν τη δουλειά τους ή την καριέρα τους, γιατί συχνά δεν έχουν αυτή την αίσθηση του στόχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, κύριε Ισλερ. η κυρία Κοράτσα Μπίλτ από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων της ε, Γυναίκας και της Ότας των, των Φίλων δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας για λόγους απρόβλεπτους. Ξεκινούμε λοιπόν τη συζήτηση. Αλλά ξεκινώντας θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έχει ετοιμάσει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μικροεκθέσεις για την ισότητα των γυναικών. Ο τίτλος είναι ο εξής. Γυναίκα, ούτε, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Και εδώ έχουμε ακριβώς την ευκαιρία να συστήσουμε αυτή την σύντομη έκθεση. Μετάβαση από το 19ο στον 20ο 21ο αιώνα. Η γιαγιά μου δεν μπόρεσε να μάθει να διαβάζει για να μην ε, πάμε τα μυαλά της αέρα. Η μάνα μου δεν μπόρεσε να τελειώσει το, το μεταπτυχιακό της γιατί θεωρήθηκε ότι αφού τα αδέλφια της δεν μπορούσαν, δεν θέλανε να σπουδάσουν, δεν θέλανε να πάνε στο πανεπιστήμιο, δεν έπρεπε και εκείνη να κάνει κάτι παραπάνω από τα γόρια της οικογένειας. Εγώ μπορεί να μην έχω εγγονή τώρα, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτά τα σύνορα και αυτά τα όρια. Eh. Έχω αρκετά εκτενή κατάλογο και μια και έχουμε μια κάποια καθυστέρηση θα ακούσουμε πέντε παρεμβάσεις και μετά αναλόγως θα προσπαθούμε να δεχόμαστε τις ε, ομιλίες στα ε, επόμενα θέματα. Δύο λεπτά η κάθε παρέμβαση. Μάρτα Ματράη. Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, όταν μιλούμε για γυναίκες και αγώνες για τα δικαιώματά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιτυχία μπορούμε να έχουμε μόνο εάν αγωνιστούμε όλοι μαζί. Και αν εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα για εκπαίδευση για τους πάντες. Αυτό σημαίνει χειραφέτηση για τον πολίτη, δυνατότητα να αναπτυχθεί, να επιλέξει. Η πολιτική στην Ουγγαρία εστιάζεται στο να προσφέρει στις γυναίκες ε, την ευκαιρία και να μορφώνονται και να δουλεύουν και να κρατάνε την οικογένειά τους στο σπίτι και να τη φροντίζουν. Ισότητα υπάρχει φυσικά με τους άντρες, προβλέπεται άλλωστε και στο σύνταγμά μας και ιδιαίτερα προστατεύουμε το, τα άτομα με αναυπηρίες ή άλλες ομάδες μειονεκτικές. Οι γυναίκες χρειάζονται τη μεγαλύτερη χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη όταν θέλουν να σπουδάσουν, όταν θέλουν να βρουν μια θέση εργασία. Και εκεί θέλει η κυβέρνηση να τις βοηθήσει. Επί παραδείγματι, μια γυναίκα που έχει ένα παιδί μικρό, έχει πιο ευνοϊκέ συνθήκε για να ξεκινήσει ανώτατε σπουδέ, ε, χρηματοδότηση, υποστήριξη με υποτροφίε κτλ. προβλέπονται και άλλα μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών που θέλουν να σπουδάζουν μεγαλώνοντας ταυτόχρονα τα παιδιά τους. Η Ουγγρική κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για να ενισχύσει την ε, ισότιμη μεταχείριση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και χαιρετίζω όλους, όλες και όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ειρήνη Μαυρονικόλα από την Κυπριακή Βουλή. Είναι μέλος της ε, Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών. Έχετε το λόγο κυρία Μαυρονικόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε κυρία Πρόεδρε. Να πω ότι τα στερεότυπα κοινοτροπίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στις αναπτυγμένες και στις υποανάπτυκτες. Στην Κύπρο, ναι, έχουμε πρόβλημα με τα στερεότυπα και τις νοοτροπίες, όπως σε πολλές άλλες χώρες. Εκείνο το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών. Να μεταδώσουν σωστά το μήνυμα της ισότητας στα παιδιά να τους μεταδώσουν το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν καλύτερα σε θετικές επιστήμες και άνθρωποι που μπορούν καλύτερα σε πρακτικές επιστήμες. Ότι το τι επιλέγεις να σπουδάσεις δεν έχει να κάνει με το φύλλο, δεν έχει καμία σχέση με το φύλλο αλλά με το μυαλό. Στην Κύπρο γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε μια επιτροπή προώθησης της ισότητας στα σχολεία. Και έγινε μόλις πρόσφατα αυτό. Αντιλαμβανόμενοι ακριβώς αυτή την ανάγκη, γιατί στην πατρίδα μας όταν δείτε αποτελέσματα προεισαγωγικών εξετάσεων, οι γυναίκες παίρνουν πάντα τις πρώτες δέκα θέσεις και μετά εξαφανίζονται. Μόλις τελειώσουν το πανεπιστήμιο, ξαφνικά εξαφανίζονται. Δεν συμμετέχουν πουθενά. Γιατί, γιατί ακριβώς θεωρούνται ότι ε, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουν είναι να μείνουν στο σπίτι ή το πολύ το πολύ να εργαστούν αλλά να εργαστούν ως έναν ορισμένο επίπεδο. Εκείνο το οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι να, να γίνουν σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς στα παιδιά αλλά και στους γονιούς. Και είναι αυτός ο στόχος ο οποίος έχουμε μέχρι το 2018 το οποίο νομίζουμε είναι σημαντικό ακριβώς για να αλλάξει την νοοτροπία και τα στερεότυπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και ε, της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Γιούτο. Σας ευχαριστώ. Σήμερα γιορτάζουμε μια πολύ σημαντική μέρα που μας θυμίζει όλες τις σημαντικές επιτυχίες που έχουν ε, καταφέρει μέχρι τώρα οι γυναίκες αλλά και μας ε, επιτρέπει να σκεφτούμε πόσο δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε. Η παιδεία είναι σίγουρα ένα στοιχείο κλειδί έτσι ώστε η γυναίκα να μπορεί να είναι απόλυτα ο εαυτό τη και να μπορεί να επιβεβαιωθεί στο πολιτιστικό και στον επαγγελματικό τομέα. Ωστόσο θα πρέπει πολλά να γίνουν ώστε να πληρωθεί αυτό το κενό, το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε όλες τις ανισότητε και τι διακρίσει, α πούμε όλε οι γυναίκε και οι κοπέλε οι Ευρωπαίε, οι οποίε επιτυχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στι σπουδέ του και είναι πανέτοιμες και ικανές, είναι πραγματικά άριστες και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτές. Όμως στη συνέχεια όλες οι προσπάθειες αυτές που έχουν γίνει στα σχολεία ή στα πανεπιστήμια ε, ξανεμίζονται όταν μπουν στο χώρο, χώρο της εργασίας. Και σκέφτομαι όλα αυτά τα κορίτσια που για παράδειγμα στην Ιταλία ενώ έχουν ε, πολύ ψηλό πτυχίο έχουν ένα δίκτυο απασχόλησης πολύ χαμηλό, ιδιαίτερα στις μεσογειακές ε, στις νότιες περιοχές και εκεί που βρίσκουν απασχόληση ε, δεν είναι αντίστοιχη με τα πτυχία τους τα επαγγελματικά ούτε ε, ο μισθός που παίρνουν αντιστοιχεί στις σπουδές τους. Θα πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει και να, προ... να οθήσει τα κράτη-μέλη, να πιέσει τα κρατη ώστε να ασκήσουν πολιτικέ που θα οδηγήσουν στην υπέρβαση αυτού του προβλήματο. Ελπίζω σε ένα χρόνο να μπορούμε να ξαναμιλήσουμε εδώ και να σημειώσουμε κάποιο πρόοδο που θα έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιούτο. Εκ μέρου τη Μαλτέζικη Βουλή, το λόγο έχει η κυρία Τζοβάνα Ντεμπόνο. Ευχαριστώ πρόεδρε και καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό τοποθετείται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για να εξασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων όσο υπάρχουν ακόμη αποκλήσεις στις ευκαιρίες για την εκπαίδευση και, πάνω από, και εξίσου σημαντικό την κατάρτιση θα συνεχίσει να παραμένει το χάσμα στην ισότητα των φύλων. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου στα κράτη-μέλη και προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση και για τα δύο φύλλα. Αυτό άνοιξε νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες για ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο δεν έχει με αυτό εξαντληθεί το ζήτημα. Ε, το, ο αγώνας για την ισότητα των φύλων δεν μπορεί να σταματάει στο πανεπιστήμιο. Δεν αρκούν μόνο τα πανεπιστημιακά πτυχία και οι δεξιότητες οι θεωρητικές και δεν πρέπει να ε, ανεχόμαστε να μένουν άχρηστες ή να ξεπερνιούνται. Πρέπει να μπορεί μια γυναίκα να έχει πρόσβαση στην κατάρτιση σε όλη της τη ζωή. Δεν πρέπει μόνο να δέχεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά σε όλη τη διάρκεια του βίου της, του βίου της μέχρι και τα γυρατιά. Μόνο έτσι μπορεί να μεγιστοποιηθεί ο πολύτιμος αυτός πόρος. Πιστεύω λοιπόν ότι η έννοια της ελεύθερης κατάρτισης και της αναβάθμισης των ικανότητων για τις γυναίκες έχει τεράστια σημασία για τη συμμετοχή τους στην παραγωγική απασχόληση και τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν νέε δεξιότητες, ακόμη και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ύστερα από μία έως και ε, παρατεταμένη απουσία για οποιονδήποτε λόγο. Πιστεύω ότι πιο φιλόδοξοι στόχοι πρέπει να προσδιοριστούν λοιπόν από εδώ και μπρο και πρέπει να κάνουμε περισσότερο ώστε να ενθαρρύνουμε τι ηλικιωμένε γυναίκε στην εξασφάλιση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και άλλων ε, ε, γνώσεων που θα χρειαστούν στη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ρόλο καθοριστικό στην κοινωνία και να διατηρήσουν κάθε δυνατότητα διαφύλαξης των πνευματικών δυνατοτήτων τους ε, και του δυναμικού τους, ανεξαρτησία, ε, δυνατότητα να προσδορίζουν το μέλλον τους και βέβαια να συμβάλλουν στην ευημερία των οικογενειών και της κοινωνίας. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης, η κυρία Βέσνα Μάροβιτς έχει το λόγο. Βέσνα Μάρκοβιτς. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή μου σε αυτή τη διάσκεψη και τη δυνατότητα που μου δίνεται να λάβω το λόγο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ε, σίγουρα ε, μεγάλη πρόκληση και λύση είναι η πρόσβαση στην ε, μόρφωση. Έτσι θα χειραφετήσουμε τις γυναίκες ε, και θα τις επιτρέψουμε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Έτσι θα εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία τους ε, και την ε, λήψη ελεύθερων και τεκμηριωμένων αποφάσεων. Είναι πολύ ευαίσθητες και τις ομάδες των, γυναικών, κυρίως των, γυναικών που ζουν ε, στην Ήπεθρο ή έχουν αναπηρίες, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και δεν μπορούν να τα ασκήσουν. Ε, προσπαθούμε να, να συμπεριλάβουμε στην, στη Σερβία και τα κορίτσια σε πλήρη ε, άσκηση των δικαιωμάτων, να απαγορεύουμε την, ε, διακριτικές τη διακριτική μεταχείριση και τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Βέβαια υπάρχουν πολλές διακρίσεις εξαιτίας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ε, κοινωνικής κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να, αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, ε, να πατάξουμε την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών και φυσικά να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα. Δυστυχώς εξακολουθούν να ισχύουν τέτοια στερεότυπα σε συγκεκριμένες ομάδες όπως στους ΡΟΜ που δεν έχουν υψηλά επίπεδα φίτησης, ειδικά των κοριτσιών στα σχολεία δυστυχώς ε, ε, τέτοια, τέτοια στερεότυπα οδηγούν στην ε, περαιτέρω διάκριση εις βάρος των, των γυναικών. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε φυσικά από την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ισότητα ανδρών και γυναικών όταν διδάξουμε στα παιδιά τον αμοιβαίο σεβασμό. Ε, θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τις γυναίκες σε πιο περιθωριοποιημένες ομάδες και να εξασφαλίσουμε την, την πρόσβασή τους σε όλα τα επίπεδα της ε, παιδείας. Εμείς στη Σερβία κάνουμε προσπάθειες ε, εξασφάλισης αυτής της ισότητας. Διοργανώνουμε διασκέψεις για την αντιμετώπιση της αδικογενειακής φίας, της θέσης των γυναικών Ρωμά, της ισότητας των φύλων. Επίσης, υιοθετήσαμε την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας εις βάρος των γυναικών. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους μηχανισμούς ε, προκειμένου να εντάξουμε στην εσωτερική μας ένωμη τάξη νόμους και διατάξεις ε, που θα υλοποιήσουν αυτή την ισότητα των δύο φύλων σε, όλα τα, σε όλους τους τομείς δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του τομέα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας, την κυρία Μικαέλα Σόντροβα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω κι εγώ. Ως νεότερο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να πω όμως ότι ήμουν και στο Τσεχικό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και ως Εθνική Βουλευτής είχα εκφράσει την υποστήριξή μου στην ισότητα των φίλων για την εκπαίδευση και έχω εκφράσει την υποστήριξή μου στη ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για όλους, ώστε να μπορέσουν να ε, διεκδικήσουν το συμβασμό των δικαιωμάτων τους. Και υποστηρίζω ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση ε, το, της εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων στην Ινδία για τα, ε, μικρά, για τα κορίτσια στην Ινδία. Θυμάμαι τα ονόματα όλων αυτών των κοριτσιών που έχουμε βοηθήσει να πάνε στο σχολείο και με τα οποία ακόμα κρατάω επαφέ. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε και παιδιά έξω από την Ευρώπη. Γιατί η κατάσταση εκεί είναι συνήθως πολύ πιο δύσκολη. Σαν μήνυμα μπορώ να πω ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η κυρία Χάουα Ιμπραχήμ μας είπε ότι η εκπαίδευση ήταν αυτή που της έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις τις... τα τυχερά που της ήρθανε. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει τυχαία να συμβαίνει η εκπαίδευση. Είναι κάτι που πρέπει ενεργά να υποστηρίξουν οι κοινωνίες μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις γυναίκες και τα κορίτσια. Είναι πιο έξυπνα άλλωστε και γι' αυτό πρέπει να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που προσφέρεται να δώσουμε εκπαίδευση στα κορίτσια. Για κοιτάξτε στα πανεπιστήμια, πιο πολλά είναι τα κορίτσια που σπουδάζουν από τα γόρια... στην Ευρώπη. Γιατί οι γυναίκες έχουν ε, τη βούληση να μορφωθούν. Η μελέτη της ε, Πίζας του 2012 δείχνει ακριβώς ε, αυτή την βούληση ότι τα κορίτσια στο πανεπιστήμιο έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια. Ε, αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι καλύτερες επιδόσεις οφείλονται στην ε, φιλοδοξία, στη βούληση να έχουν καλύτερους βαθμούς και αποτελέσματα. Ωστόσο και πέραν αυτού δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι γυναίκες έχουν και έναν άλλο ρόλο. Θέλουν να είναι μητέρες, ε, να φτιάξουν μια οικογένεια. Και εδώ έρχεται η σύγκρουση μερικές φορές. Γιατί και τη δουλειά τους θέλουν να κρατήσουν, αλλά και παιδιά να κάνουν. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσει η κοινωνία, τη γυναίκα, να εξασφαλίσει την ε, λεπτή αυτή ισορροπία μεταξύ του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου και άρρωστα αυτό ισχύει και για μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Και για να ολοκληρώσουμε την πρώτη θεματική ενότητα, γιατί έπονται και άλλες δύο. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν την πρώτη θεματική ενότητα, θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπάσινη Μέτ από την Τουρκία, πρώην Υπουργό ε, Παιδείας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης ε, και είναι βουλευτής της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι συμμετέχοντες. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της ε, συνάντησης αυτής, να υποστηριχθεί για άλλη μια φορά η σημασία της εκπαίδευσης για τις γυναίκες και να δοθούν ευκαιρίες για αλλαγή. Σε κάθε τομέα της ζωής, όπου δραστηριοποιείται η γυναίκα, βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Από το 19ο αιώνα αρχίζουν οι γυναίκες να συμμετέχουν στο κοινωνικό βίο, να καταρτίζονται, να εκπαιδεύονται, να εργάζονται. Αλλά από τότε αρχίζουν και τα εμπόδια απέναντι στα οποία πρέπει να αγωνιστούν. Τώρα, η μεγάλη αλλαγή που έχει επέλθει είναι ότι τα προβλήματα των γυναικών δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. στα τελευταία 12 χρόνια στην Τουρκία βλέπουμε μια μεγάλη και ιστορική προσπάθεια για αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε να πραγματοποιήσουμε σημαντικά βήματα προσφέροντας υποστήριξη και κίνητρα. Στον αγώνα για την ε, διεκδίκηση των δικαιωμάτων της γυναίκας περιλαμβάνεται η μόρφωση αλλά και διεκδικήσεις που φτάνουν μέχρι την κατάρριψη ε, παγιωμένων ιδεών και νοοτροπιών. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Για το 2002 καταρχάς, όπου είχαμε στις εκλογές μόνο 24 γυναίκες στο, Ευρω... στο τουρκικό κοινοβούλιο, ενώ στις εκλογές του 2011 είχαμε 79 γυναίκες βουλευτές με συμμετοχή από την πρώτη φορά στο 4,4 και μετά το 14%. Βλέπουμε μια τεράστια λοιπόν αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων, στους μηχανισμούς λήψη αποφάσεων. Αυτό φέρνει και αλλαγές στις νοοτροπίες στην κοινωνία κάθε μέρα βλέπουμε ότι καταρρύπτεται και ένα εμπόδιο ή μία ε, προκατασκευασμένη ιδέα. Εμείς συνεχίζουμε αυτές τις προσπάθειες και θεωρούμε ότι πρέπει να ενταθούν ακόμη περισσότερο. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών αποτελούν ένα εμπόδιο στο να αναπτυχθεί μια κοινωνία πλούσια με ποικιλία ανοιχτή σε όλους. Κάθε είδους λοιπόν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών θα πρέπει να καταρρύπτονται, να αντιμετωπίζονται και αυτό με την ανταλλαγή απόψεων και τον διάλογο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μέσα. Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα για να εξασφαλίσουν όλα τα δικαιώματα και την ισότιμη μεταχείριση γυναίκες, δεν το αρνούμαστε αυτό. και προβλήματα τα οποία θέλουμε να υπογραμμίσουμε για να συζητηθούν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις ε, εντάσεις και τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιφερειά μας που σημαίνουν πως πολλές γυναίκες πέφτουν θύματα βίας. Έχουμε δύο εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες που έχουν αναστήσει καταφύγιο και άσυλο στην Τουρκία. Πρόκειται για έναν ε, πληθυσμό μεγάλο, ανθρώπους που δραπετεύουν από τις συνθήκες του πολέμου που επικρατούν στη Συρία. Κατά 85% από ό,τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί και ο Οργανισμός Εθνών είναι γυναίκες και παιδιά, αμόρφωτες συχνά, γυναίκες που χρειάζονται υποστήριξη αυτή τη στιγμή η Τουρκία δορίζει, διαθέτει 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των ε, προσφύγων αυτών, ε, της ε, σύντησή τους, τη στέγασή τους και ταυτόχρονα και την μόρφωση στο βαθμό που μπορούμε να προσφέρουμε. Έτσι λοιπόν και αυτές τις μέρες που μιλούμε για τα δικαιώματα των γυναικών θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα το ζήτημα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες. Σε αυτές πρέπει να προσφέρουμε μια προσέγγιση υγεία, μια προσέγγιση με όρους αλληλεγγύης. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Νιμέτ. Ξέρουμε. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, αλλά πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο μας, γιατί αν ο καθένας ή καθεμία μακρηγορεί, θα στερεί την ευκαιρία σε άλλους συναδέλφους να μιλήσουν αργότερα. Και νομίζω ότι η αυστηρή τήρηση του χρόνου είναι και ένδειξη αλληλεγγύης προς τους επόμενους ομιλητές. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να δώσουμε το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες. Περάμε τώρα στη δεύτερη θεματική ενότητα, στο δεύτερο πάνελ με θέμα της προκλήσης για μια ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Στο δεύτερο αυτό πάνελ έχουμε τρεις καλεσμένες. Θα δώσω το λόγο στην πρώτη μας ομιλήτρια, την κυρία Βίνκελε, πρώην Υπουργό Πρόνοιας της Λετωνίας και είναι μέλος ε, της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών της Βουλής της Λετωνίας. Κυρία Βίνκελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και καλημέρα σας. Βέβαια στην, ε, στην σημερινή πραγματικότητα δεν αρκεί να έχει μόνο κανείς μια δεξιότητα. Και αυτό είναι δύσκολο να το αντιληφθεί και να το συνειδητοποιήσει κανεί στι χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ συμπεριλαμβανομένη και τη Λετωνία. Κατά την Σοβιετική εποχή η ζωή ήταν πολύ απλούστερη. Το ιδανικό σενάριο ήταν το εξή. Γύρω στην ηλικία των 22-23 ετών ε, αποφυτούσαμε και μετά εργαζόμασταν ε, μέχρι την σύνταξή μας ε, στον τομέα στον οποίο είχαμε σπουδάσει και οι γυναίκες συνταξιδοτούνταν γύρω στα 55. Σήμερα η ποιότητα της ε, παιδείας ε, αποδεικνύεται όχι μόνο από πτυχία ε, έγκυρων πανεπιστημίων, αλλά καθορίζεται και από την προσαρμοστικότητα του καθενός στην μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη αγορά εργασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λετωνία δίνουν έμφαση στην οικονομία της γνώσης και γι' αυτό χρειαζόμαστε ειδικού στις τεχνολογίες. Σε πολλές χώρες και στη Λετωνία οι άνδρες δεν συμμετέχουν ιδιαίτερως στην οικογενειακή ζωή. Οπότε οι γυναίκες δεν έχουν ισότιμες ευκαιρίες με τους άνδρες εκτός της οικογενειακής ζωής. Υπάρχει άνηση σχετικά κατανομή των ευθυνών και αυτό οφείλεται κυρίως σε ισχυρά στερεότυπα για τους παραδοσιακούς ρόλους ε, των ανδρών και των γυναικών. Ε, στερεότυπα που ισχύουν όχι μόνο στην ιδιωτική ζωή αλλά και στην επαγγελματική ζωή. Τα στερεότυπα εξαρτώνται από τη, την κοσμοθεωρία και το σύστημα των αξιών και των αρχών. Και φυσικά η νοοτροπία δεν αλλάζει μόνο δια νόμου. Τα στερεότυπα οδηγούν ε, σε διακρίσεις μεταξύ των φύλων και στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Οι γυναίκες της Λετωνίας έχουν συγκριτικά ε, καλύτερη μόρφωση από τους άντρες, αλλά εκπροσωπούνται πολύ λιγότερα στις τεχνολογίες που είναι κινητήρια μοχλή της οικονομίας και επίσης δεν εκπροσωπούνται ιδιαίτερο στην αγορά εργασίας. Μόνο το 20,6% των πτυχιούχων από τεχνολογικά προγράμματα είναι γυναίκες. Ενώ οι γυναίκες πτυχιούχοι στις οικαστικές τέχνες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στις ιατρικές επιστήμες είναι περίπου 90%. Πολλά προβλήματα παρεμποδίζουν την ε, ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στη διαβίω κατάρτιση. Επειδή ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες προσχολικής εκπαίδευσης και βερφονιπιακών σταθμών, οι γυναίκες αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Οπότε έχουν λιγότερες ευκαιρίες να συνεχίσουν την μόρφωσή τους, να επιστρέψουν στην αγροναργασία ή να ολοκληρώσουν τις σπουδέ τους. Μόνο οι νέοι ε, ε, ε, αξιοποιούν τέτοιες ευκαιρίες και κυρίως όσοι είναι ειδικευμένοι. Όσοι είναι ανειδίκευτοι έχουν ακόμη λιγότερες ε, πιθανότητες να συνεχίσουν τις σπουδέ τους. Επίσης οι γυναίκες δεν παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως γιατί δεν μπορούν να συμφιλιώσουν την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική. Και τέτοια τους προγράμματα προσαρμόζονται στις, αγορές, στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δηλαδή επικεντρώνονται σε τεχνικές δεξιότητες ε, που θεωρούνται κατά παράδοση ανδρικό προνόμιο. Η Λετωνία είναι μικρή χώρα και στην έκταση και στον πληθυσμό. Η πρόσβαση όμως ε, δυστυχώς ε, στη διαβίου κατάρτιση είναι άνηση μεταξύ ανδρών και γυναικών και στις αρακοτικημένες περιοχές η ανισότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ούτε η εξαποστάσεως ε, μάθηση προωθείται ιδιαίτερος. Και η διαβίου κατάρτιση είναι δαπανηρή, γιατί προϋποθέτει ε, μεταφορά από το χώρο διαμονής στο χώρο φίτησης, κάτι που δεν μπορούν να το ε, πληρώσουν όλοι. Επίσης, οι γυναίκες σε ηλικία προσυνταξιοδότησης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να, να μην βρουν ε, θέση απασχόλησης όταν την έχουν χάσει. Θα πρέπει λοιπόν ε, να στηρίξουμε τους εργοδότες, ε, να, προσλαμβάνουν υπαλλήλους από τέτοιες ομάδες. Ε, δεν υπάρχουν και αρκετά κίνητρα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την έναρξη νέας σταδιοδρομίας και την παραμονή στην αγορά εργασίας και είναι δαπανηρές αυτές οι διαδικασίες, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις δημοτικές ή εθνικές αρχές. Παροχές δηλαδή συμβουλών ε, επαγγελματικού προσανατολισμού. Βέβαια τέτοιες προκλήσεις ε, δεν είναι μόνο ε, πρόβλημα της Λετωνίας. Αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες μέλη παρόμοια προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε από κοινού τις καλύτερες λύσεις. Εν κατακλείδη θα ήθελα να σας αναφέρω και ένα θετικό παράδειγμα από τη Λετωνία. Για πέμπτη συνέχεια χρόνια η, η επιχείρηση τηλεπικοινωνιών που είναι κατά το ίμιση κρατική διδάσκει δεξιότητες χρήση υπολογιστή σε ηλικιωμένους Μάλιστα η μεγαλύτερη μαθήτρια ήταν 90 ετών, γυναίκα. Και ο συνολικός αριθμός των ηλικιωμένων που σπουδάζουν τέτοιου είδους υπολογιστές μάλλον από αυτό το πρόγραμμα είναι γύρω στους 10.000. Thank you. Ε, Σας ευχαριστώ. Το, δεύτερο, το λόγο έχει τώρα η κυρία Ρεμπέλο που είναι πρόεδρος του ε, πορτογαλικού δημοκρατικού κινήματος γυναικών και το θέμα είναι η ίση ισότιμη παιδεία. Οι γυναίκες ανέκαθεν αγωνίζονταν για τα δικαιώματά τους ε, ε, παράλληλα με τους άντρες. Όμως στην Πορτογαλία το 1974 αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και τότε ε, άρθηκαν όλες οι διακρίσεις που βασίζονταν στο φύλλο και επέτρεπε έτσι ότι στις γυναίκες η πρόσβαση στην παιδεία, στην ενημέρωση, στο στη κουλτούρα, σε όλες τις θέσεις ε, και που αλλιότερα ήταν απαγορευμένα. Ε, το Πορτογαλικό Σύνταγμα θεωρεί την ισότητα ως βασική του αρχή και εγγυάται ότι όλοι οι πολίτες έχουν την ίδια κοινωνική κατάσταση και είναι ε, ίσοι απέναντι στον νόμο. Δικαίωμα λοιπόν στην παιδεία και στη βασική παιδεία. Οι κοπέλες μπορούσαν λοιπόν να μπουν στη σύστημα το εκπαιδευτικό χωρίς εμπόδια ε, και αυτή η κατάσταση έχει διαρκώς βελτιωθεί στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών. Ταυτόχρονα με την έλευση της δημοκρατίας στην Πορτογαλία το 1985 ε, καθιερώθηκε το διεθνές, ε, ε, η Διεθνής ημέρα μάλλον για τις γυναίκες και γίναν διάφορες διάσκεψεις και σύνοδοι μέχρι ότου που φτάσαμε στο 1995 στην τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες όπου παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα πρόγραμμα δράσης ε, που εστιαζόταν σε δύο βασικούς τομείς ε, την βιώσιμη ε, ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης αλλά και των ευκαιριών για τα δύο φύλλα. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τη διάσκεψη του Ποκίνου και επιβάλλεται να ρωτήσουμε. Καταρχήν, έχουν ε, υλοποιηθεί οι στρατηγικοί στόχοι της πλατφόρμας δράσης, ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό τομέα όσον αφορά την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, την πρόσβαση στο σχολείο και το επίπεδο των προσόντων τους. Και δεύτερον, αν λάβουμε υπόψη τις ε, κοινωνικές και οικονομικές αλλά και τις πολιτικές αλλαγές που έχουν συμβεί στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, χρόνια ποια είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων και γενικότερα στην κατάσταση της γυναίκας. Στη χώρα μας το 2002 35% των κοριτσιών ανάμεσα στα 20 και τα 24 έτη είχαν ε, τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην ανώτατη εκπαίδευση 65% είναι γυναίκες και σε όλους τους τομείς της γνώσης. Η παρουσία η γυναικεία είναι μεγάλη στη, στην παιδεία γενικότερα και φτάνει στο 81% και στο τομέα των μηχανικών φτάνει στο 30% οι γυναίκες ε, επιδιώκουν περισσότερο τη συνέχιση των σπουδών τους. Το 2012, 54,2% των Πορτογαλίδων είχαν, ε, πάρει το, είχαν πετύχει στο πτυχίο τους και παρά τις διάφορες μελέτες που γίνονται και που επιβεβαιώνουν την επιτυχία των γυναικών στις σπουδές, υπάρχει διαρκώς μια διάκριση και μια υποβάθμιση των γυναικών στην χώρα της εργασίας τους. Και σας δώσω κάποια παραδείγματα. Όσον αφορά τους καθηγητές και τους δάσκαλους, πιο πολύ εκεί είναι η μεγάλη η παρουσία. Όμως όταν φτάσουμε στους καθηγητές και αυξάνεται μάλλον το επίπεδο της εκπαίδευσης, μειώνεται και η συμμετοχή των γυναικών. Φτάνουμε στο 44% όταν φτάνουμε στους καθηγητές πανεπιστημίων με την ίδια πτυχία και τις ίδιες, ε, τα ίδια προσόντα στους διαγωνισμούς όσον αφορά την επιτυχία των υποψηφίων ε, συστηματικά επιλέγονται οι γυναίκες. Το ίδιο και στις πανεπιστημιακές έδρες όπου είναι μεγαλύτερες οι δυσκολίες για τις γυναίκες. Εδώ το ποσοστό στα δημόσια πανεπιστήμια ε, συμμετοχής των γυναικών είναι μόλις 22%. Στην έρευνα οι γυναίκες διακρίνονται σε όλες ε, τους τομείς σπουδών στην ιατρική, στις, ε, στην ε, αγρονομία, στη παρουσία τους είναι λίγο λιγότερη ε, στο τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας. Σε σχέση με τον τομέα όπου ασκούν τις δραστηριότητες μου, βλέπουμε ότι 2 εκατομμύρια αντιστοιχούν στο Ε, στα 2 εκατομμύρια μάλλον θέσεις απασχόλησης έχουμε 61% γυναίκες και 30% άνδρες. Οι άνδρες ωστόσο κατέχουν τις ψηλότερες θέσεις. Αυτές οι διαφορές μας δίνουν τις, ε, ε, τα δεδομένα αλλά και τις προκαταλήψεις που ισχύουν απέναντι στις γυναίκες. Εξακολουθεί η γυναίκα να θεωρείται η μόνη υπεύθυνη για τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας αλλά και της φροντίδας για την εκπαίδευση των παιδιών. Ενώ εργάζεται και εκείνη το ίδιο. Στον ερευνητικό τομέα οι γυναίκες είναι πολύ φιλόδοξες και εφευρετικές και πολύ συχνά λαμβάνουν βραβεία για τις ανακαλύψεις τους ή τις εφευρέσεις τους. Πρόσφατα μάλιστα ε, στην εφαρμοσμένη βιολογία ήταν γυναίκα εκείνη που κέρδισε το βραβείο. Έχουμε πολλά υποσχόμενες γυναίκες, αλλά δυστυχώς οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται περισσότερο. Η διεθνή επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιολογηθεί η γυναικεία προσπάθεια. Δεν αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο το εκπαιδευτικό σύστημα επέτρεψε να αναγνωριστούν οι ικανότητες, τα προσόντα και οι γνώσεις ε, και οι δεξιότητες των γυναικών, αλλά και μάλιστα οι επιτυχίες τους πολλές φορές είναι μεγαλύτερες από το, αυτές των ανδρών. Όμως η συμμετοχή στην κοινωνική, στην επαγγελματική και στην οικονομική ζωή δεν είναι ισότιμη και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να προωθηθεί η ισότητα της σταδιοδρομίας στα πανεπιστήμια, στα Ινστιτούτα, στα Ιδρύματα, στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι το δημοκρατικό σχολείο είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να προωθήσει την ε, ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Η δε κρίση οικονομική επέτεινε πτυχές που είναι πραγματικά ε, ε οπισθοδρομικές. θα πρέπει το υλικό, το παιδαγωγικό να προσαρμοστεί. Δεν έχει τελείως αφαιρεθεί από εκεί η σεξιστική εικόνα για τις διάφορες, τα διάφορα επαγγέλματα. Και επίσης παρουσιάζονται οι γυναίκες με τρόπο παραδοσιακό ας πούμε. Ε, περιλαμβάνονται επίσης τάσεις και παρεμβάσεις των καθηγητών, των δασκάλων, των γονέων που θα πρέπει να προτείνουν διαφορετικές δραστηριότητες ε, για τις ε, κοπέλες, για τις γυναίκες. Οι κοπέλες πολλές φορές στα κορίτσια έχουν πολλές περισσότερες ικανότητες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων μαθημάτων. Και αυτή τη διαφορά θα πρέπει, θα πρέπει να τη θεωρούμε φυσική. Η στάση αυτή τελικά μπορεί να οδηγήσει στην ε, ε, συμπεριφορά αυτή των καθηγητών. Μόλις περάσαμε σε ένα καινούριο αιώνα θα πρέπει να κρατήσει ισότητα για όλους, ε, να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θα πρέπει ε, ωστόσο μέσα σε αυτή την κρίση την οικονομική και την πολιτική να προσέξουμε γιατί εμφισβητούνται τα δικαιώματα που έχουν επιτευχθεί. Μέχρι στιγμής τα αρνητικά, οι αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα της παιδείας ε, επιβιώνονται από σχετική έρευνα που έγινε το 2014. Στη χώρα μας οι πολιτικές ε, λιτότητας των τελευταίων κυβερνήσεων επηρέασαν πολύ σημαντικά το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η Πορτογαλία, ο πεδίο είναι και λιγότερο σε αυτό το θεμελιώδη τομέα για την ανάπτυξη και αποδίδει μόλις 3,6% του ΑΕΠ του, του ΑΕΠ της, κάτω δηλαδή από το μέσο όρο του ΩΣΑ που είναι 3,25. Επίσης πανούμε πολύ λιγότερα για την κατάρτιση πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. 200 εκατομμύρια ευρώ θα αφιερωθούν το 2015 στην δημόσια εκπαίδευση και έτσι επηρεάζεται η λειτουργία ε, και η ε, εξωσχολική παιδεία γενικότερα. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Πορτογαλία δεν ε, συνδέονται με κανένα σχέδιο υπέρ της ισότητας η βασική εκπαίδευση έχει οδηγηθεί σε υποβάθμιση, έχουν μειωθεί οι απαιτήσει, έχει απαξιωθεί το καθεστώς των καθηγητών, είναι ασταθής η ζωή στη ζωή, ε, είναι συγκεκριμένες περιστάσεις που επηρεάζουν και το εναρχή της ισότητας της παιδείας για τα κορίτσια και για τα αγόρια, όπου αυτό καθιερώνεται στο Σύνταγμά μας. Θα πρέπει λοιπόν να εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε για τη συγκεκριμενοποίηση των στόχων της πλατφόρμας του Πεκίνου. Οι απαραίτητε επενδύσει από τι κυβερνήσει θα πρέπει να γίνονται για την εκπαίδευση, να αυξάνεται η ποιότητα και η ισότητα των ευκαιριών για του άνδρες και τι γυναίκε, για όλες τους τομείς της γνώσης. Επίσης η προώθηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου όπου τα κορίτσια θα ενθαρρύνονται να ασχολούνται με διάφορα πεδία γνώσης ώστε να διευρύνουν τις ευκαιρίες τους για την μελλοντική τους σταδιοδρομία, να εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε για μια, ένα κοινοτικό σχολείο το οποίο αξιοποιεί τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις καθώς και να υπάρχει ένας χώρος για τον πολίτη όπου τα κορίτσια με τα γόρια συνεργάζονται και μοιράζονται τις ευθύνες, που, πράγμα που τους προετοιμάζει για μια πραγματική συμμετοχή ισότιμη σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρεμπέλο. Τελευταία ομιλήτρια της δεύτερης ε, θεματικής ενότητας είναι η κυρία Αγνιέσκα Κοσλόφσκα, μέλος της Επιτροπής Γυναικών, θα μας μιλήσει για τις ε, ευρωπαϊκές προκλήσεις ε, παραθέτοντας και τις εμπειρίες της από την ε, εποχή που θύτευσε ως υπουργό Ίσης Μεταχείρισης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τα πρώτα λεπτά της παρουσίασής μου να σας μιλήσω για την κατάσταση ισότητας των δύο φύλων και μετά να μιλήσω για την παιδεία. Το θέμα της ισότητας των δύο φύλων το αντιμετωπίζουμε σε τέσσερις βασικούς τομείς που έχουν θεμελιώδη σημασία. Είναι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών που προσκρούει στο μισθολογικό χάσμα και στο συνταξιοδοτικό χάσμα. Είναι πραγματικά απογοητευτικοί οι δείκτες και είναι χαρακτηριστική της ε, έλλειψης που έχουμε σε κάποια κράτη-μέλη της ισότητας των δύο φύλων. Δεύτερο δεύτερος σημαντικός τομέας είναι η δυνατότητα παράλληλης υλοποίησης των ε, στόχων στην οικογενειακή ζωή και στον επαγγελματικό βίο. Τη συμφιλίωση δηλαδή της οικογενειακής ζωής, ε, της μητρότητας με την επαγγελματική εξέλιξη. Τρίτος τομέας σημαντικός είναι η παρουσία των γυναικών στη, σε, θέσεις ε, διευθυντικές, ηγετικέ ε, στη συμμετοχή ε, στη λήψη αποφάσεων. Και εδώ είναι σημαντικά τα πολιτιστικά δυστυχώ στερεότυπα που ίσχυε μερικέ φορέ και εμποδίζουν τι γυναίκε να προσχωρήσουν σε αυτέ τι ηγετικέ θέσει. Και σημαντικό άλλο τομέα είναι η βία. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο τομέα, το μισθολογικό χάσμα που είναι 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, ενώ το συνταξιοδοτικό χάσμα είναι 39% στις διαφορές γυναικείων ανδρικών συντάξεων. Δηλαδή, η μέση κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε ε, μήνα λαμβάνει σύνταξη που είναι κατά 40% χαμηλότερη από ε, ανδρική σύνταξη. Κάτι που δείχνει τις διαφορές, την ανισότητα, τα εμπόδια των πολιτικών μας. Και είναι σημαντικός αυτός ο τομέας της ε, οικονομικής εξάρτησης των γυναικών της κλίμακας ε, ένδυας των γυναικών. Και μάλιστα τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε δεν λαμβάνουν πολλές φορές υπόψη τις άνεργες γυναίκες. Τις γυναίκες ε, που δεν έχουν ούτε δικαίωμα σε σύνταξη, ούτε λαμβάνουν κάποια κοινωνικά επιδόματα. Οπότε είναι ακόμη μεγαλύτερη η φτώχεια των γυναικών, γιατί στο μέσο όρο δεν λαμβάνονται τέτοιες κατηγορίες γυναικών υπόψη. Ένα άλλο τομέα που σας είπα είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης ε, υλοποίηση των προσωπικών και των επαγγελματικών στόχων. Μιλούμε για το δικαίωμα των γυναικών ε, στην απασχόληση. Ναι, σίγουρα υπάρχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, παρόλο που μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση, αλλά το δύσκολο είναι η υλοποίηση ε, του στόχου τη μητρότητα, του προσωπικού στόχου τη αυτοεκπλήρωσης μέσω τη μητρότητα. Γιατί δεν είναι ελεύθερη επιλογή να γίνει κάποια γυναίκα μητέρα και μετά να επιδιώξει και επαγγελματική σταδιοδρομία. Με ελάχιστε εξαιρέσει, όλες οι γυναίκες οφείλουν να εργαστούν και έχουν ανάγκη να εργαστούν. Δεν μπορούν απλώς να κάθονται σπίτι και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Οπότε έχει νόημα ε, ο αγώνας των σύγχρονων φεμινιστριών υπέρ της ίσης πρόσβασης. Ενώ οι γυναίκες, πολύ, οι άνδρες, συγγνώμη, πολύ εύκολα και χωρίς κανένα πρόβλημα μπορούν να συμφιλιώσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Και μάλιστα οι άνδρες που έχουν παιδιά ευνοούνται στην αγορά εργασίας. Αυτό δείχνουν οι μελέτες. Ενώ τα παιδιά και η οικογένεια είναι βάρος στις γυναίκες που θέλουν να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία. Είναι πρόβλημα και όταν θέλουν να συνεχίσουν και να επανέλθουν στην αγορά εργασίας μετά τη μητρότητα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά, γι' αυτό και χρειάζεται σημαντική κοινωνική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα προωθεί στην ισότητα των δύο φύλων. Υπάρχουν φοβερές δυσαναλογίες και στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και επίσης μεγάλη δυσαναλογία στον, στον επιμερισμό των ευθυνών εντός του, σπιτιού, του νοικοκυριού. Η μέση γυναίκα ε, εργάζεται 49 44 ε, ε, ώρες την εβδομάδα, ενώ 41 ο άνδρας, ενώ η γυναίκα στη δουλειά, ενώ στο σπίτι 39 ώρες η γυναίκα και 8 ώρες ο άνδρας στο σπίτι. Υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία, μεγάλες διαφορές στο χρόνο εργασίας και στη δουλειά και στο σπίτι μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες γενικώ ε, ε, δουλεύουν πολύ περισσότερο. Εννέα ώρες τη βδομάδα μία γυναίκα δουλεύει περισσότερο από έναν άντρα. Και μάλιστα οι γυναίκες ε, έχουν τριπλάσιο αριθμό ορών απλήρωτων. Κάτι που δημιουργεί μεγάλες ανισότητες και προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Και αυτές οι διαφορές σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στα στερεότυπα και στις κοινωνικέ κοινωνικές πολιτικές. Θα πρέπει να προωθήσουμε μια πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών και στο σπίτι μεταξύ των ανδρών και γυναικών. Γιατί έχουμε τα στερεότυπα της χιονάτης, της ταχτοπούτας, ε, είναι γυναίκες που περιμένουν τον πρίγκιπα να τις απελευθερώσει, να τις σώσει. Αυτά είναι στερεότυπα και δυστυχώς ε, συνοδεύουν τη ζωή πολλών γυναικών σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες. Θα πρέπει αυτά τα στερεότυπα να τα καταρρύψουμε χάρη στην μόρφωση, χάρη στην εκπαίδευση. Και ερχόμαστε στο θέμα της εκπαίδευσης. Πολύ σωστά επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα της εκπαίδευσης, γιατί από ποσοτική άποψη έχουμε υλοποιήσει τους στόχους. Η ποιότητα είναι που μας διαφεύγει προς το παρόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή των γυναικών στην παιδεία, στην συνέχιση των σπουδών, στην ε, επαγγελματική κατάρτιση, εκεί πολύ συχνά, συχνότερα οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε παιδεία σε σχέση με τους άντρες. Και οι επενδύσεις ε, που κάνουν οι γυναίκες στην παιδεία δεν πιάνουν τόσο τόπο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της θέσης απασχόλησης ε, ε, όσο οι αντίστοιχες επενδύσεις που γίνονται στους άνδρες. Παρόλο που οι γυναίκες ε, σπουδάζουν πολύ περισσότερα από ό,τι οι άνδρες και παρακολουθούν και επαγγελματική κατάρτιση, δεν βελτιώνεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Οπότε έτσι χάνουμε τα ταλέντα μας κατασπαταλούμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που συσσωρεύουν οι γυναίκες στη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ προωθούμε περισσότερο τα ταλέντα και τις δεξιότητες των ανδρών, αφήνοντας αναξιοποίητο το δυναμικό των γυναικών. Θα πρέπει να διορθώσουμε λοιπόν αυτές τις ανισότητες και αυτό θα πρέπει να γίνει όσο, όχι μόνο μέσω της επίσημης ε, της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και της ανεπίσημης, με μέντορη, με παροχή συμβουλών, με αλλαγή της νοοτροπίας και της διαπαιδαγώγησης και στην αγορά εργασίας και όχι μόνο στα σχολεία. Σε ό,τι αφορά την επίσημη εκπαίδευση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που αναφέραμε και εδώ, στο θέμα των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των ε, πολιτιστικών ε, ιδεών που μας οδηγούν ε, να μεταχειριζόμαστε διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες. Και μερικέ φορέ οι επιλογέ στη σταδιοδρομία οφείλονται ακριβώ στην άνηση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση ακόμη και στην προσχολική ηλικία. Γιατί ακόμη και εκεί τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Βλέπουμε κούκλες μόνο και κάποια βαρετά παιχνίδια για τις γυναίκες, ενώ πολύ περισσότερα παιχνίδια για τα αγόρια. Και μάλιστα ε, επιτέλους πριν από χρόνια διαβάσαμε ότι η Lego έβγαλε ε, φιγούρες ε, τεχνικών, μηχανικών που επιτέλους δεν έχουν μόνο ανδρική μορφή αλλά περιέλαβε και τις γυναίκες στα, η Lego στα σχέδιά της. Είναι σημαντικό λοιπόν να αλλάξουν τα στερεότητα ακόμη και στη, στα παιχνίδια. Θα πρέπει να επιτρέψουμε και να ανοίξουμε κάποιες τεχνολογίες ε, και κάποιους τομείς περισσότερο και στις γυναίκες, γιατί οι διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή οφείλονται περισσότερο στα στερεότυπα. Επίσης, ε, τα κορίτσια και μετά οι γυναίκες, ακόμη και στη λογοτεχνία, είναι ηρωίδες ε, σε μειονεκτική θέση, παθητικές. Αυτή, αυτά τα στερεότυπα επηρεάζουν ε, την αντίληψη που δημιουργούμε στη συνέχεια για τους παραδοσιακούς ρόλους των ανδρών και γυναικών. Και τα σχολικά βιβλία είναι σημαντικό στομέας. Πολλές φορές, ακόμη και στα σχολικά βιβλία, διονίζονται αυτά τα στερεότυπα και οι παραδοσιακοί ρόλοι. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Δεν θα πρέπει τα σχολικά βιβλία να διαιωνίζουν τα στερεότυπα. Και τα, βλέπουμε τέτοια στερεότυπα και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, για παράδειγμα, οι ανδρικές και οι γυναικείες φιγούρες είναι τελείως διαφορετικές. Για παράδειγμα, οι άνδρες είναι ε, θαραλέοι ήρωες, γενναίοι, ενώ οι γυναίκες ε, έχουν ε, ίσονα σημασία ρόλους, είτε είναι υπηρέτριες, είτε είναι μητέρες, είτε σύζυγοι. Ελάχιστα ε, έχουμε παρουσία γυναικών στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως σούπερ ηρωίδων με υπερφυσικές δυνάμεις. Περισσότερο άνδρες έχουν αυτούς τους ρόλους, ακόμη και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και κάτι από την προσωπική μου ζωή. Πριν από λίγο καιρό ήρθε 7χρονος γιος μου στο σπίτι και μου είπε επιτέλους ε, έχουμε μια φεμινιστική, ε, φεμινιστική αλλαγή στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μπορούμε να δούμε και γυναίκες, γυναικές μορφές ε, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και σε σημαντικούς ρόλους. Οπότε τα στερεότυπα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σημαντικά και το θέμα της, ε, το επικίνδυνο φαινόμενο της ε, ε, σεξουαλικής παρουσίασης των γυναικών μέσω των διαφημίσεων, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι γυναίκες προ... παρουσιάζονται σεξουαλικό ενδικήμενο. Αυτό επηρεάζει με πολύ αρνητικό τρόπο και πολύ επικίνδυνο τρόπο την διαπαιδαγώγηση. Και μερικές φορές διονύζει την ανισότητα. Λοιπόν, συνοψίζοντας, σημαντική είναι η ποιότητα της παιδείας, η ποιότητα της μόρφωσης, ε, λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των δύο φύλων και την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης ε, εξαιτίας του διονυσμού των στερεοτύπων που δυστυχώς ε, εξακολουθούν να υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις τρεις ε, καλεσμένες της δεύτερης θεματικής ενότητας για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που μας έκαναν και που σίγουρα δημιούργησαν τροφή για σκέψη, όπως θα φανεί και στην ε, ακόλουθη συζήτηση. Επιμένω και σας θέλω παρακαλώ να σεβαστείτε το δίλεπτο στις ομιλίες σας. Πρώτος ο κύριος Ζεράρ Κρόουλη, πολύ φοβάμαι ότι κατακρεούργησα στην προφορά το επώνυμό σας. Είναι μέλος ε, της Επιτροπής ε, ε, Πρόνοιας και Παιδείας της Γερουσίας της Ισλανδίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κρόκουελ. Ζερόμ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο του καθηγητή της επαγγελματικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού και γενικότερα των ε, δασκάλων και των γονιών. Ο καθηγητής της, του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει κρίσιμο ρόλο. Μπορεί να καθοδηγήσει κορίτσια όπως και αγόρια στην επιλογή μη τετριμένων, μη συμβατικών ε, σταδιοδρομιών. Και έτσι πρέπει ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση σε αυτό το θέμα. οι οδηγοί ε, επαγγελματικού προσανατολισμού λοιπόν έχουν μπει στην Ιρλανδία ε, στο σύστημα το σχολικό ε, δικέ διοικητικά, ξαναμπήκανε μέσα στις τάξεις και πρέπει να περάσουμε πλέον όχι μόνο σε μια ουδέτερη στάση απέναντι στα φύλλα, αλλά πρέπει να περάσουμε στη συνειδητοποίηση ότι ο καθένα μπορεί να είναι επηρεασμένο ω προ τη θέση των φύλων, ιδιαίτερα οι γονεί. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε προ μια δραστήρια ε, αλλαγή θεώρηση. Ε, εάν ε, ρωτήσετε έναν άντρα τι θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει στη ζωή της μια γυναίκα, εγώ Φερρυπίν που έχω δύο μικρές αδελφές, γυναίκα και κόρη, ε, θα σας απαντήσω το ίδιο πράγμα που θα ήθελα να κάνουν και τα αγόρια της οικογένειας. Αυτό θα σήμαινε πραγματική ισότητα στη θεώρηση των φίλων. Στην ε, Ιρλανδία πρέπει πιστεύω να πούμε ότι χρειάζεται να προβληθούν και οι τεχνολογίες και οι σταδιοδρομίες που, έχουν, που βγαίνουν από τα παραδοσιακά και, και την πεπατεμένη. Πρέπει να βοηθήσουμε και άλλα κορίτσια, ε, όχι μόνο τα ολίγα, τις ολίγες εξαιρέσεις, να βγουν από το καλούπι της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Το Code Dojo που είδαμε, το, πρόγραμμα εξοικείωσης με τους υπολογιστές και τον προγραμματισμό, του οποίου ένα παράδειγμα είδαμε νωρίτερα με ένα κορίτσι που μας μίλησε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και θέλω επίσης να πω ότι εάν δεν κάνουμε τίποτα άλλο, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μία λύση μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα εντοπίζει τον πρωταθλητή της ισότητας σε κάθε σχολείο, κοινωνία, κοινότητα που θα προάγει αυτήν ακριβώς την ιδέα. Η Αμερικανίδα ομιλήτρια νωρίτερα για να ολοκληρώσω είπε ότι διστάζουμε να μιλήσουμε για φίλο. Ε, κοιτάξτε, πριν να παντρευτώ, για το σεξ μάλλον, πριν να παντρευτώ, ξέρετε, την παραμονή του γάμου μου, μου με πιάνει η μητέρα μου και μου λέει ε, αγόρι μου πρέπει να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό και εγώ της είπα ας το μάνα σε έχουν ξεπεράσει εξελίξεις αυτά και ευχαριστώ Muchas Σας ευχαριστώ από την Κροατική Βουλή τώρα, το λόγο έχει η κυρία Ντούνα Εσπολιάρ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα σχολεία στην ε, ε, Κροατία δυστυχώς ε, διονύζουν τα στερεότυπα. παρουσιάζονται τα γόρια ως επιμελή εργατικά, θαραλέα, ενώ γυναίκες ως τρυφερές, ωραίες, αλληλέγγυες. Έχουμε περισσότερο τις γυναίκες στο ρόλο του θύματος και του, αγοριού στο ρόλο του, του ήρωα και του σωτήρα. Ε, τα αγόρια εκπαιδεύονται να γίνουν πιλότοι και οι γυναίκες και τα κορίτσια δασκάλες. Οπότε πολύ πιο σπάνια έχουμε τις γυναίκες ως συγγραφείς. Έχουμε περισσότερο στο ρόλο, ε, στην λογοτεχνία τις γυναίκες στο ρόλο των γυναικών, των συζύγων και, και πολλές φορές και στην ύπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε το ρόλο των γυναικών στην, ε, στην οικογένεια, γιατί δυστυχώς ε, αυτό είναι το στερεότυπο, ότι οι γυναίκε ασχολούνται με το νοικοκυριό, με το σπίτι, ανατρέφουν τα παιδιά και πολύ σπάνια τις βλέπουμε στην αγορά εργασία. Και όταν τις βλέπουμε εκεί τότε είναι είτε νοσοκόμε, είτε δασκάλε, είτε πολίτριες. Και είναι καυγαδε... οι γυναίκε ε, ευερέθιστε, καυγατζούδε ε, και δειλές. Ενώ οι άντρες είναι ηγέτες, αποφασιστικοί, θαραλέοι και οι εξισώσεις στην Κροατία είναι γυναίκα ίσως σπίτι, ε, άντρας δουλειά. Πώς θα αλλάξουμε λοιπόν αυτή την οτροπία. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολικά βιβλία, να, να αποφύγουμε την, ε, ε, παραδοσιακή παρουσίαση των στερεοτύπων ρόλων. Επίσης, ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μία μεταρρύθμιση που έχει ήδη ξεκινήσει του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να εκπαιδευτούν οι ε, καθηγητές ε, στην ισότητα των δύο φύλων και να αποφύγουν ε, διπλά μέτρα και σταθμά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Επίσης, με τα σχολικά βιβλία και την σωστή αγωγή του πολίτη να προωθήσουμε, θα προωθήσουμε την ισότητα των, των δύο φύλων θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση των διδασκάλων. Θα πρέπει επίσης ε, να λάβουμε υπόψη ότι την, το προηγούμενο μήνα αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο στην Κροατική Βουλή, οπότε ε, από τις επόμενες ε, εκλογές θα έχουμε ποσόστοση γυναικεία τους ε, στα εκλογικά ψηφοδέλτια με συμμετοχή 40% των γυναικών. Αλλιώ, δεν θα νομιμοποιείτε ακόμα να κατέβει σε εκλογέ αν δεν εξασφαλίσει αυτή την ποσόστοση. Σα ευχαριστώ. Εκ μέρου τη πορτογαλική βουλή τώρα, το λόγο έχει η κυρία Έτσα Πάη. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματο του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου θα ήθελα να χαιρετήσω το Ευρωκοινοβούλιο για αυτή την πρωτοβουλία και να ε, συγχαρώ την κυρία Ρεβέλο που αντιπροσωπεύει μία από τις παλιότερες μη κυβερνητικέ οργανώσεις της Πορτογαλίας. Θα ήθελα να, εστιάσω, να ξεκινήσω τη δική μου ε, παρέμβαση παραθέτοντας την Μαλάουα που πήρε το το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και το βραβείο Σαχάροφ που είπε ότι η παιδεία είναι τα πάντα για τα κορίτσια. Είναι τα πάντα για τα κορίτσια στην Ασία, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και γι' αυτό θα πρέπει να φωτίσουμε και να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα περί φύλου που έχουν εμποδίσει από τις γυναίκες και τους άντρες να έχουν μία ζωή, μία οικογένεια με ισότητα ευκαιριών. Έχουν περάσει, έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα. Ένα μεγάλο κομμάτι των, της διαδρομίας ε, στην ιατρική αλλά και στην ε, κοιοσύνη είναι γυναίκες, ενώ άλλοι τομείς κυριαρχούνται από τους άντρες. Χρειαζόμαστε ωστόσο μια παιδεία για την ηθαγένεια ε, σε αυτή ε, της επικράτειας της Ευρωπαϊκής και αυτό προχωράει στην Πορτογαλία αλλά και στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε κοινωνικές πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε με τα στερεότυπα και να προωθήσουμε την ε, συμφιλίωση ανάμεσα στην εργασιακή και στην οικογενειακή ζωή. Όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες. Γιατί οι, άντρες, οι γυναίκες έχουν πολλές δυσκολίες ε, να ε, κάνουν διαδρομία, αλλά και οι άντρες αντίστοιχα έχουν, πρέπει να οθηθούν να συμμετέχουν περισσότερο στις οικογένειές τους γιατί έτσι θα είναι ο κόσμος πιο ίσος, πιο δίκαιος θα υπάρχει ισότητα ευκαιριών ε, ανεξάρτητα από το φιολογικό τους φύλλο με το οποίο γεννιούνται οι άντρες και οι γυναίκες. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα έχει το λόγο εξ ονόματος του Ευρωκοινοβουλίου η κυρία Σνεγέρ Πιέρης. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zit hier nu en ik dacht aan 30 jaar geleden. 30... Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάθαμε εδώ και σκέφτομαι τι γινόταν πριν από 30 χρόνια όταν ήμουν στην Ολλανδία, δεν είχα μορφωθεί, ήμουν γεωργός και ήθελα να μπω στην πολιτική και να δραστηριοποιηθώ και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ακολουθήσω μαθήματα για την ε, ε, μαθήματα ρητορικής ε, ήταν πολύ ακριβά μαθήματα, αλλά μου προσέφεραν πάρα πολλά ε, όσον αφορά την στήριξή μου, γιατί μπορούσα έτσι να πω ε, τι πίστευα και έτσι οι άνδρες που βρίσκονταν κοντά μου άρχισαν να με σέβονται και άρχισα να επισκέφτομαι οργανώσεις των γυναικών που ήταν πολύ ισχυρέ στις κατοχώρες και έλεγαν πόσο σημαντικό ήταν να δραστηριοποιηθεί κανείς στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις. 30 χρόνια μετά επιστρέφω Ευρωκοινοβούλιο ενώ πίστευα ότι έπρεπε σχεδόν να συνταξιδοτηθώ, αλλά μετά επανήλθα και πέτυχα 130.000 ψήφους. Και αυτό δεν ήταν μόνο από γυναίκες αυτές οι ψήφοι, και πολύ συχνά βλέπω πως οι γυναίκες ε, ζηλεύουν η μια την άλλη, δεν στηρίζουν πάντοτε η μια την άλλη. Είναι σημαντικό ωστόσο να έχουμε την ε, γυναικεία στήριξη και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε γιατί οι άντρες έχουν ε, καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις και το έχω κάνει αυτό συστηματικά. Πολύ συχνά μπορεί κανείς να προσελκύσει τους άντρες ε, ε, στις δικές του πεπιθήσεις. Έχω και εγώ δύο κόρες που είναι στον τομέα των μέσων μαζική ενημέρωση, αλλά πρέπει να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τι γυναίκε ώστε να ξεπεράσουν τα πρώτα εμπόδια στην μόρφωσή του. Σα ευχαριστώ. Ε, το στις Bundestag τη Γερμανία, η κυρία Δωροθέα Τέλε. Σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τη Γερμανία, το σπίτι. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι η αλλαγή των ε, ρόλων, των παραδοσιακών ρόλων, μπορεί να γίνει και μέσω των ασομαζικής ενημέρωσης. Ε, έχουμε παραδείγματι τελευταία εξασφαλίσει την υποστήριξη και για τον ελάχιστο μισθό που είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις γυναίκες και την ε, ε, ενίσχυση, το επίδομα που παίρνουν οι γυναίκες όταν μένουν στο σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ε, για ένα χρόνο. Έχουμε εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες μετά τη γέννηση ενός παιδιού και αύριο ψηφίζεται η αύξηση στο 30% του, της ποσόστοσης για τη συμμετοχή των γυναικών στις σταδιοδρομίες κτλ. Είναι όπως υπόθηκε νωρίτερα, αναγκαίο να αλλάξουμε την εικόνα της γυναίκας. Χρειαζόμαστε γυναίκες στο ρόλο του προτύπου και στη δικτύωση, όπως έχουν κάνει οι άντρες εδώ και αιώνες. Πρέπει να δικτυώνονται οι γυναίκες και να υποστηρίζουν οι γυναίκες. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 7.4 της προτάσεως για τα σχολεία ε, μόνο θηλεών ή μόνο αρένων ε, και σε μία μελέτη που έχω κάνει ε, χρόνια τώρα που δείχνουν ε, πόσο πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα προσφέρουν σχολές ή σχολεία που ασχολούνται μόνο με κορίτσια ή μόνο με αγόρια και κυρίως στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολύ συχνά μετά τα 12-13 κυρίως τα κορίτσια, οι πιο μικρά ακόμα μπορεί να, είναι, να παίζουν το ρόλο της ταχτοπούτας, της χιονάτης, να ονειρεύονται πώ θα είναι και αργότερα μπάρμπι. Ε, αυτό λοιπόν το παραδοσιακό, τον παραδοσιακό ρόλο των γυναικών πρέπει να τον ανατρέψουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ελληνικό Κοινοβούλιο τώρα. Η κυρία Φωτεινινάκη. Ah. Thank you very much, Chair. Um, I come from... Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Είμαι Ελληνίδα. Πριν εκλεγώ στο Κοινοβούλιο ήμουν ε, πανεπιστημιακός και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που απορρέουν από τη δική μου εμπειρία στο Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό που ονομάζεται κατάρτιση εκπαιδευτικών, εκπαίδευση εκπαιδευτικών δασκάλων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα πρέπει να είναι σε θέση να, να δώσουν κατευθύνσεις ε, και νοοτροπία ουδέτερη προς το φύλλο γιατί μόνο με τους προσανατολισμούς και την εκπαίδευση μπορεί να απελευθερωθεί, να χειραφετηθεί το ανθρώπινο μυαλό, να διαραγούν τα πρότυπα και να αλλάξει η ιστορία. Τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια βλέπουμε ευτυχώς θετική εξέλιξη, εξέλιξη ως προς την, ε, τις μελέτες για το φύλλο, κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες γίνονται πιο πολλά μαθήματα, αλλά και έργα, project, που χρηματοδοτούνται για τις μελέτες τις σχετικές με την ισότητα των φίλων, την ηθαγένεια, την συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και τη δημοκρατία. Και τώρα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να βγω, να βγω λίγο από το θέμα αυτό για να αναφερθώ στην πρακτική υλοποίηση. Παρά το ότι υπάρχει η ισότητα των φίλων στην ελληνική εκπαίδευση ως αρχή, μεγάλη είναι η απόκληση που διαπιστώνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση, στον επαγγελματικό χώρο και δεν αναφέρομαι τόσο σεξουαλική παρενόχληση όσο στην, ε, στις διακρίσεις προς τις δυνατότητες απασχόλησης ανάλογα με τα φύλλα πρώτο θύμα της τεράστιας οικονομικής κρίσης ήταν οι γυναίκες. Οι πρώτες οι οποίες επιλέγησαν για, επιλέγονται για ευέλικτη μερική απασχόληση ήταν οι γυναίκες. Οι γυναίκες ήταν και αυτές που πρώτες απολύονται ή αποκλείονται για λόγους εγκυμοσύνης ή μητρότητας. Σε, σε θέσεις υψηλού κινδύνου γυναίκα δεν, παίρνουν, δεν προσλαμβάνουν γιατί δεν έχει δικαίωμα να είναι μητέρα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σας ευχαριστώ. Muchas gracias. Ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα της ε, Επιτροπής ε, Εργασία Απασχόλησης της ε, Σουηδικής Βουλής Το λόγο έχει ο συνάδελφος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ θερμά για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της διάσκεψης. Στη... Οι γυναίκες ανέκαθεν έχουν μικρότερη εκπροσώπηση στην πολιτική σε σχέση με τους άντρες και από τη στιγμή που ισχύει αυτό το φαινόμενο, καθώ και το φαινόμενο τη ενδοοικογενειακή ε, βία ή τη βία κατά των γυναικών, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, είμαι υπερήφανο γιατί στη Σουηδία έχουμε φεμινιστή πρωθυπουργό. Μάλιστα είναι και μέλος της ε, οργάνωσης που αγωνίζεται για την εξασφάλιση της ισότητας. Έχουμε φεμινιστική κυβέρνηση, φεμινιστές ε, υπουργούς που δίνουν μάχη για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων. Και το κυβερνητικό έργο είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε εξασφάλιση της ισότητας. Έχουμε σχεδόν πλήρη ισότητα σε πολιτικό επίπεδο και θέλουμε να τη μεταφέρουμε και στον εργασιακό χώρο. Γιατί αν θέλουμε μία ίση κοινωνία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε απασχόληση και να μειώσουμε τις διακρίσεις. Βέβαια, δυστυχώς, ούτε και στη Σουηδία έχει εξασφαλιστεί πλήρης ε, ισότητα, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που περισσότερο ε, μένουν στο σπίτι και ανατρέφουν τα παιδιά τους ε, και έχουν τις περισσότερες δουλειές άνευ αποδοχών ή φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς. Δεν είναι άντρες που αναλαμβάνουν τέτοιες υποχρεώσεις. Οπότε θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας ε, και τώρα και στο μέλλον, ώστε κάποια στιγμή να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ισότητα των δύο φύλων ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο των δυναμικών και των ανδρών και των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κος. Τώρα από τη Μαλτέζικη Βουλή το λόγο έχει η κυρία Μαρλέν Φερούκα. Πρόεδρε, όπως πολλοί το έχουν αναφέρει, αλλά και η Μανών το τόνισε στην δική της ε, παρουσίαση, ζούμε σε μια εποχή όπου οι νέοι διδάσκουν τους πιο Επίσης ζούμε σε μια εποχή όπου η παιδεία και ο τρόπος που διαβιβάζεται στους δυνητικούς ε, σπουδαστές κάθε ηλικίας έχει ε, πάρει νέα μορφή. Γιατί, Γιατί όταν ήμασταν νέοι μας έλεγε η κοινότητά μας, η κοινωνία μας, η οικογένειά μας, το σχολείο μας να μας μάθαινε. Τώρα μας διδάσκουν οι κοινωνίες, οι οικογένειές μας, τα σχολεία μας, αλλά και τα κοινωνικά, τα μέσα μάλλον κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η, η κυβερνοεκπαίδευση, η οποία μπορεί να είναι κρίσιμη, όπως πιστεύω, στην κάλυψη των χασμάτων, των κενών που υπάρχουν ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν πρόσβαση στην παιδεία και εκείνες που δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία. Άλλη μου παρατήρηση είναι ότι βρισκόμαστε εδώ γιατί θέλουμε να έχουμε γυναίκες ευτυχισμένες και ε, που έχουν υλοποιήσει τα όνειρά τους και ε, άντρες ε, που έχουν υλοποιήσει τα όνειρά τους και είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και για να γίνει αυτό είναι ισότητα, ίσες ευκαιρίες είναι πολύ σημαντικές αλλά για να μπορούμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις άντρες και στις γυναίκες τις ευαισθησίες των γυναικών ή των ανδρών να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαφορές διαφορές στη ζωή μιας γυναίκας έτσι ώστε αυτές οι διαφορές να μην εμποδίζουν την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Muchas gracias. Continuamos eh, con el debate intentando incorporar. Συνεχίζουμε. Προσπαθώ να δώσω το λόγο και σε ομιλητές που είχαν ξεμείνει από τον προηγούμενο γύρο. Η κυρία Σουσάνα Ρος από, το, από την Ισπανική Βουλή. Ευχαριστώ. Ο Νέλσον Μαντέλα είπε ότι η μόρφωση, η παιδεία είναι το σημαντικότερο όπλο για να αλλάξουμε τον κόσμο. Και η επένδυση στην παιδική ηλικία μέσω της παιδείας είναι η καλύτερη επένδυση και σημαντική ε, αλλαγή για τις κοινωνίες ε, και για τα άτομα, για, τις, για τα παιδιά και για, ε, τα κορίτσια. Κανένας δεν μπορεί να στερήσει, να αφαιρέσει κανείς γνώσεις που έχουν εσωματωθεί. Είναι σημαντικό όπλο και για να καταπολεμήσουμε την βία. Θα πρέπει να διδαχθούμε την αρμονική και ισότιμη συνύπαρξη. Μόνο με τη μόρφωση θα καταπολεμήσουμε την ανισότητα και η καλύτερη μόρφωση και η καλύτερη παιδεία είναι αυτή που, δίνεται ισότιμα στα αγόρια και τα κορίτσια. Επίση, η παιδεία θα πρέπει να αποκλεί κανέναν. Ε, μιλήσαμε για συνεκπαίδευση, με ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το δικαίωμα κάθε κορίτσι και κάθε γυναίκα, να απολαύσει τι ευκαιρίε τα δικαιώματα, να μην βιώσει βία και να ακούγεται τη φωνή τη στην κοινωνία, όλα αυτά θα απειληθούν αν το κορίτσι ή η γυναίκα δεν μπορεί να πάει σχολείο να σπουδάσει. Όταν ένα κορίτσι πηγαίνει στο σχολείο, αναπτύσσει τι γνώσει και τι δεξιότητε τη, θα μπορέσει να λάβει πιο τεκμηρωμένε αποφάσει και πιο ελεύθερε στην ενήλικη ζωή. Θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, ελεύθεροι, σίγουροι και χειραφετημένοι. Η μη ε, κυβερνητική οργάνωση Plan International ε, μιλάει για την αύξηση κατά 20% των ε, αποδοχών ε, για τα κορίτσια που σπουδάζουν. Και φυσικά αυτά, αυτή η αύξηση των αποδοχών θα επενδυθεί στην κοινωνία. Δεν θα πρέπει να παλιδρομήσουμε ούτε στα δικαιώματα στην παιδεία, στα δικαιώματα των παιδιών, στην ανάπτυξη και στη γνώση. Η επένδυση στη μόρφωση των κοριτσιών είναι από τις πιο έξυπνες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση θα ενισχύσει το εργατικό δυναμικό, τις δεξιότητες και θα αυξήσει και το ΕΠ. Και τέλος ήθελα να πω ότι η ισότιμη εκπαίδευση δεν είναι μόνο αυτός σκοπός, αλλά ο δρόμος για την ουσιαστική δημοκρατία, για την ανάπτυξη και για την οικονομική ανάταξη των χωρών μας. Η καλύτερη επένδυση μιας χώρας είναι η επένδυση που γίνεται στην παιδεία. Ευχαριστώ. Eh. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα από την Ιταλική Βουλή το λόγο έχει η κυρία Μάρα Καρότσι. Σας ευχαριστώ. Στη χώρα μου καταγράφουμε πολλές πρόοδους ε, στην ε, ε, στην παρακολούθηση των σχολείων από τα κορίτσια αλλά και σε, στην ανώτατη εκπαίδευση συμμετέχουν περισσότερα κορίτσια. Όμως τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε δει ότι τα κορίτσια είναι χειρότερα στα επιστημονικά θέματα, από ότι τα αισθητικές επιστήμες από ότι τα χωριά και αυτό είναι γιατί συνήθως ε, ε, αντιμετωπίζουν ε, με πολλούς, ε, πολλή ενέργεια και πόρους ε, το άγχος τους αντί να αφιερώνουν αυτή την ενέργεια στην μάθηση. Για να ξεπεραστεί αυτό το θέμα νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαν πολλοί, να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα τα οποία επιμένουν και γι' αυτό κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 ε, ίσες ευκαιρίε για όλους ε, ε, συμμετείχαν εκεί όλοι για να μπορέσουμε ακριβώς να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα. Δυστυχώς με τα χρόνια εγκαταλείφθηκε αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα, αλλά τα στερεότυπα όχι και καθορίζουν τις επιλογές των παιδιών, των αγοριών και των κοριτσιών. Γι' αυτό προσπαθούμε να ξαναρχίσουμε τη δουλειά πάνω σε αυτά τα θέματα, ευαισθητοποιώντας τους εκδοτικούς οίκους αλλά και τους Εκπαιδευτικού ούτω ώστε τουλάχιστον στο σχολείο να ξεπεραστούν τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υφίστανται. Πιστεύω πως υπάρχουν πιθανότητε για επιτυχία, γιατί έχουν αυξηθεί πολύ οι ε, βουλευτίνες στο κοινοβούλιο μα σε σχέση με παλιότερα και για πρώτη φορά οι γυναίκες είναι το 1 τρίτο του κοινοβουλίου μα. Σα ευχαριστώ. Muchas gracias. Ε, Ευχαριστούμε. Από τη Βουλή του Κωσυφοπεδίου το λόγο έχει η κυρία Άλμα Λάμα. Uh, thank you. I'll speak in Albanian. Ε, ευχαριστώ, θα μιλήσω αλβανικά. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές των άλλων εθνικών, των εθνικών κοινοβουλίων, πιστεύω, θα ήθελα από πράγματα που ήδη σε μεγάλο βαθμό έχουν καλυφθεί. Η κατάσταση που έχουμε στην ε, χώρα μου μοιάζει πολύ με αυτά που βλέπουμε σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση στα παιδιά τους δίνουν οι δάσκαλοι και μάλιστα οι δασκάλες. Οι δασκάλες είναι αυτές οι οποίες ε, διδάσκουν τα παιδιά, αλλά με σχολικά βιβλία που έχουν γράψει άντρες. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξαλείψουμε τη διάκριση και την εικόνα της διαφοράς μεταξύ των φίλων; Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φεμινιστής ή φεμινίστρια για να αντιληφθεί ότι αυτή η νοοτροπία περνάει μέσα από όλες τις εικόνες και τα μηνύματα των σχολικών βιβλίων για τον παραδοσιακό ρόλο των φίλων που παρουσιάζουν τα κορίτσια Φερρυπίν να, κάνουν, να αναλαμβάνουν δραστηριότητες ε, λιγότερο σημαντικές ή δύσκολες, λιγότερο δύσκολες από ό,τι τα αγόρια. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας, η κάθε χώρα, να επενδύσει στην κατάρτιση των δασκάλων. Αυτοί έχουν ρόλο κρίσιμο να διαδραματίσουν. Και βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε την αναφορά της ε, ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης ε, μέσα στις ίδιες τις οικογένειες. Αλλά οπωσδήποτε ο δάσκαλος πρέπει να καταρτιστεί, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί, πρέπει να εκπαιδευτεί και γι' αυτό χρειάζονται χρήματα. Πολλέ από τι χώρε τη περιοχή μα τουλάχιστον δεν διαθέτουν αρκετού πόρου για τέτοια θέματα. Και γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό οι υπουργοί παιδεία να συντάσσουν τα προγράμματά τους λαμβάνοντας υπόψη την γυναίκα και την ισότητα, αλλά και τους εκπαιδευτικούς γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ και για να ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος συζητήσεων, για να περάσουμε στην ε, επόμενη, στον επόμενο γύρο, θα λάβει το λόγο εκ μέρου ε, του Κοινοβουλίου του, της Σερβίας η κυρία Μπογδάνα Κόρμικ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι και εγώ ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργανώνει τη διάσκεψη αυτή. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πολιτική πρέπει να στρέφεται στον άνθρωπο. Στον 21ο αιώνα, την εποχή της υψηλής τεχνολογίας, της μόρφωσης, το να παραμένει κανείς αδαής θα πρέπει να είναι επιλογή. Αλλά επιλογή σημαίνει ότι έχει απόλυτη δυνατότητα πρόσβασης ισότιμα στη γνώση, την παιδεία. Και μετά να αποφασίσει να μην τη χρησιμοποιήσει αυτή την πρόσβαση. Δυστυχώς όμως από όσα ακούμε εδώ σήμερα, βλέπουμε ότι οι άνδρες στα παιδιά έχουν απόλυτη πρόσβαση, ενώ αντίστοιχα δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στα κορίτσια. Τρεις λόγους εντοπίζω εγώ για το φαινόμενο αυτό. Καταρχάς γιατί από την αρχή ανέκαθεν τις αποφάσεις έπαιρναν οι άνδρες και προσδόριζαν τους κανόνες. Για να εξασφαλιστεί λοιπόν η πρόσβαση των κοριτσιών στην ε, ύψη της ποιότητας εκπαίδευσης, εκπαίδευση, θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Θα πρέπει να έρθουν τέτοιου είδους αλλαγές που δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστούν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση. Δεύτερος λόγος. Ε, το αφήγημα για την γυναίκα που συμπεριφέρεται σωστά. Ξέρουμε τι σημαίνει να είναι μια γυναίκα αποδεκτή κοινωνικά. Δεν μπορεί να είναι μηχανολόγος, δεν μπορεί να είναι φυσικός. Εγώ, επί παραδείγματι, έχω ακολουθήσει σπουδέ φυσικού, κατά τύχη έγινα πολιτικός. Αλλά θεωρείται ότι δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό μια γυναίκα γιατί δεν είναι κομψό ε, δεν, είναι, δεν της χάρη. Ε, αυτό, τη μόρφωση και την τεχνολογία για τη γυναίκα πρέπει να την αναγνωρίσουμε ως τη νέα χάρη του 21ου αιώνα. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτό το φαινόμενο. Και τρίτος λόγος είναι ότι σε περίοδους κρίσεως, όχι μόνο οικονομικής αλλά και αξιών, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε το τίμημα της κρίσεως αυτής να το πληρώνουν τα κορίτσια και οι γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Thank you. We finish this, this panel. Ευχαριστώ. Τελειώνει εδώ αυτό ο γύρος συζητήσεων. Και τώρα για να αναλάβει την καθοδήγηση του επόμενου κομματιού και τη συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε στη χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνω τον λόγο στη συνάδελφο Σίλβια Κώστα, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Παρακαλώ, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα με μια κάποια καθυστέρηση, αλλά ήμουνα σε ένα άλλο κτίριο για άλλη διάσκεψη, πάλι εδώ στι Βρυξέλλε. που πάλι αναφερόταν σε μια πτυχή συναφή κατάρτιση και εκπαίδευση πάλι, δηλαδή τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή των Γυναικών αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή. Έχουμε μια ισχυρή ομάδα διευθυντική εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που επέλεξε αυτό το θέμα για τη σημαντική ημέρα της γυναίκας του 2015 και ξέρουμε επίσης ε, ότι η προσεχής Επιτροπή των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών έχει προσδιορίσει το θέμα αυτό ως προτεραιότητα. Για να είμαι πιο σαφής και να καταλαβαίνετε αυτά που σας λέω, αλλά και για να μπορώ να μιλάω πιο γρήγορα θα συνεχίσω στα Ιταλικά, εάν μου επιτρέπετε. Αναγνωρίζοντα ταυτόχρονα και την αρχή τη πολυγλωσία και του σεβασμού σε όλε τι κουλτούρε που έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Συνεχίζω λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω την ε, εισαγωγή σε αυτή την ε, συζήτηση, σε αυτό το κομμάτι και το γύρο των συζητήσεων με τους ομιλητές μας, τρεις τον αριθμό ύψης της ποιότητας για, και να κάνω κάποια σχόλια. Μπορεί να μην είμαι το ίδιο ειδική στα θέματα αυτά, αλλά έχουμε την κυρία Ροντρίγκες εδώ που θα λάβει το λόγο μετά για να μας μιλήσει. Θα ήθελα να πω ωστόσο, και φαντάζομαι ότι ήδη το έχετε υπογραμμίσει και εσείς, ότι Η ειρηνική επανάσταση του 19ου αιώνα ήταν η δυνατότητα για τα κορίτσια να σπουδάζουν, να πηγαίνουν στο σχολείο και να σπουδάσουν. Αντίστοιχα, στο δεύτερο κομμάτι του. Στο πρώτο, αυτό ήταν του 20ου αιώνα η επανάσταση, στο πρώτο ημίση. Στο δεύτερο ημίση του 20ου αιώνα βλέπουμε μια άλλη ειρηνική επανάσταση, ότι γίνονται οι γυναίκε ε, διδάσκαλοι. Και έτσι ανατρέπεται η επικράτηση των ανδρών, επικυριαρχία των ανδρών στον χώρο της εκπαίδευσης. Και τώρα, με το σχεδιασμό του, της Ευρώπης 2020, ορίζονται στόχοι που σε ένα βαθμό οι γυναίκες φοιτήτριες έχουν εξασφαλίσει. Ένα ζήτημα, παραδείγματι, είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την εγκατάλειψη των σχολείων σε πρώιμη ηλικία, όπου είναι 13% τα κορίτσια, ενώ 17% των αγοριών αφήνουν το σχολείο νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Και αντίστοιχα σε ορισμένες χώρες ε, τα κορίτσια είναι μόνο 12%. Ε, αυτό αναφέρεται όχι μόνο σε χώρες ε, του Βορρά προηγμένες και με χειραφέτηση αλλά και σε χώρες άλλες όπως η Μάλτα, η Ρουμανία και η Ιρλανδία. Στα πανεπιστήμια τα παιδιά του 20% ε, φοιτούν σε μεγαλύτερα ποσοστά κορίτσια στην ηλικία των 20% από αγόρια και είναι περισσότερα και τα κορίτσια που παίρνουν το πτυχίο. 40% κορίτσια. Και 60%, 60 συνολικά τα κορίτσια παίρνουν πτυχίο, ενώ είναι 40% τα αγόρια. Επίσης, βλέπουμε να παραμένουν κάποιες ε, πρώιμες διακρίσεις, σε πρώιμη φάση διακρίσεις και καθοδήγηση με βάση το φύλλο στις σπουδέ, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη, γιατί υπάρχουν παραδείγματι πολλές γυναίκες ε, στις ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά πολύ λιγότερες τεχνολογικές και τις θετικές είναι λιγότερη ενθάρρυνση που προσφέρεται στις γυναίκες ε, στο ρόλο του ερευνητή της ερευνήτριας, παρότι έχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Το ίδιο και στις τεχνικές επαγγελματικές σπουδέ και τις λοιπές δεξιότητες που θεωρούνται καθοριστικές σήμερα και απαραίτητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεξιότητες που έχουν να κάνουν με, την, ε, με τις γνώσεις και τις σπουδές στην ενέργεια, το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία. Χαμηλό είναι επίσης το επίπεδο των νεαρών γυναικών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό και νομίζω ότι πρέπει να διαρωτηθούμε και με μεγάλο αριθμό γυναικών εκπαιδευτικών που έχουμε στο, στα σχολεία μας, στην Ιταλία παραδείγματι, είναι συντριπτικά τα νούμερα υπέρ των γυναικών εκπαιδευτικών, οι οποίες μπορεί να έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά με ένα, αλλά ίσως δεν έχει φέρει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε ως προς τον περιορισμό των στερεοτύπων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των κοριτσιών, την ε, συνειδητοποίηση των ίσων ευκαιριών για τα κορίτσια και, μια, και για μια ουδέτερη προσέγγιση ως προς τις ευκαιρίες και τις προοπτικές για ε, προσωπική ανάδειξη που θα έπρεπε να ενθαρρύνονται. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Εμείς, σε παραδείγματι, στην Επιτροπή Πολιτισμού ιδιαίτερο μέλημα έχουμε την ενίσχυση των πολιτικών εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα προσέγγιση και την ε, ευαισθητοποίηση στις, ε, και την ενημέρωση ούτως των ε, εκπαιδευτικών στα θέματα αυτά. Βλέπουμε ταυτόχρονα τα κορίτσια ως υποκείμενα είναι και θύματα των διακρίσεων. Πολιτικές ε, ενσωμάτωσης, δια, διαθρησκιακό ή διομολογικό στην Ευρώπη, το πρότυπο της Ευρώπης, δείχνουν ε, και με το φως και κάποιων τραγωδιών που διαπιστώνονται σε ορισμένα κράτη, ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το ποιο σήμερα, να έρθουμε σε αντιπαράθεση με το ποιο είναι το φαινόμενο αυτό της διαπολιτισμικότητας, όχι του διαπολιτισμικού περιβάλλοντος όπως τα λέγαμε, αλλά της διαπολιτισμικότητας, τι μπορεί να προσφέρει, γιατί η γυναίκα μπορεί να προσφέρει και να πει πολλά, αφού είναι η ίδια θύμα αυτής της εσφαλμένης κουλτούρας και των διακρίσεων. Είναι σημαντικό επίσης ε, η προσεχής Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα 20 χρόνια μετά τη διάσκεψη του, Πεκίνου για την ενσωμάτωση των γυναικών, την επιλογή αυτή, την ε, στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις γυναίκες αλλά και για όλη την κοινωνία και μια εκστρατεία που έχει ξεκινήσει και ο Ομπάμα με την σύζυγό του, την Μισελ, στο, ίδιο αυτό θέμα, για να αναπτυχθούν εταιρικέ σχέσεις και με τρίτε χώρες ε, σε αναπτυξιακή πολιτική, γιατί ξέρετε εμείς έχουμε αναπτύξει μια νέα φιλοσοφία της εταιρική σχέσης, το more for more όπως λέμε, το δεύτερο more, το δεύτερο περισσότερο, το να προσφέρουμε περισσότερα για περισσότερα που θα εξασφαλίζονται, θα ήταν τα περισσότερα αυτά περισσότερη προστασία από τις διακρίσεις και περισσότερη εκπαίδευση για τις γυναίκες το δεύτερο μόρο. Επίσης ε, στην εκπαίδευση των κοριτσιών ε, ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή και για την βελτίωση των ε, συνθήκων δημόσιας οικίας, των στοιχείων και στατιστικών δημόσιας οικίας, παιδικής, μάλλον εφηβικής εγκυμοσύνης, θνησιμότητας και το καθεξής. Όλα αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε ιδιαίτερα και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα μια διάκριση η οποία δεν σημαίνει διαχωρισμό αλλά ενημέρωση ως πολιτιστική διαδικασία που περνάει μέσα από τη γνώση και που μπορεί να συμβάλλει στην εκπαίδευση. Μια γραμμική προσέγγιση είναι η εκπαίδευση η οποία συμπεριλαμβάνει και συνεπιφέρει την κληρονομιά των αξιών, της ταυτότητας, της πολιτιστικής παρακαταθήκης και αποτελεί μια πρώτη διάσταση ατομική και μια δεύτερη πιο κοινωνική διότι ξεπερνάει η εκπαίδευση τα όρια του Χολικού συστήματος, αυτό που συζητήθηκε σήμερα, ότι και μέσα και έξω από το σχολείο πρέπει να αναπτυχθούν τα λεγόμενα soft skills, οι ήπιες δεξιότητες, τις ε, ε, ηθαγένειες συμμετοχή του πολίτη, τη συμμετοχή στα κοινά, τις συνεργασίες μέσα σε μια ομάδα. Όλα αυτά που είναι τόσο σημαντικά για την ε, αλληλεπίδραση με τον άλλον και πολύ πιο σημαντικά ακόμη και από τις τυπικέ δεξιότητες που προσφέρει η εκπαίδευση. Αυτό το οποίο ξέρω πολύ καλά ότι θα αναφέρει και η ομιλήτριά μας εδώ, που αποτελούν αποτελούν τις άτυπες λεγόμενες δεξιότητες που όμως έχουν ύψιστη αξία και είναι υποχρέωση για τις αρχές των κρατών μελών να αναγνωρίζουν στο ε, σχολικό σύστημα και την εκπαίδευση, την ενίσχυση αυτών των συγκεκριμένων δεξιοτήτων όπου θα έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη οι γυναίκες και καλύτερη θέση γιατί είναι αυτή η ιδιαίτερη ε, το ιδιαίτερό τους πλεονέκτημα στην κοινωνική ε, στις κοινωνικές δεξιότητες που έχουν στρατηγική σημασία. Και έτσι νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε σε τρεις ε, κατευθύνσεις για να κλείσω. Ένα επίπεδο το οποίο θα αφορά τα πρότυπα, τα εκπαιδευτικά συστήματα μέχρι το τέλος της παιδικής ηλικίας για αγόρια και κορίτσια. Εγώ δεν είμαι υπέρ ενό συστήματος που θα λέγει ότι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε, ξέρω ότι βέβαια μεταξύ μας ε, συζητούμε χάρη στον πλουραλισμό που μας προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, όμως πρέπει να σημειώσω ότι δεν μπορούμε να λέμε μόνο ότι πρέπει να έχουμε μια ουδέτερη προσέγγιση. Εμείς έχουμε βγει όλοι από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θεωρούσε ότι ήταν ουδέτερο. Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα ότι λησμονούμε πως θα πρέπει το σχολικό σύστημα να βοηθάει το αγόρι ή το κορίτσι να αναπτύξει μια προσωπικότητα από με, αποδοχή, με αυτοπεποίθηση, με αξιοποίηση των διαφορών του, με ενίσχυση της ε, συμμετοχής του στο κοινωνικό γίγνεστη και της αυτοπεποίθησής του. Είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα και επίσης πιστεύω στον χώρο της παιδείας επίσης θα πρέπει να επανεξεταστούν διαφορετικά ψηφιακά συστήματα γιατί έχει αλλάξει πια η κατάσταση ριζικά το περιβάλλον το ψηφιακό και αλλάζουν οι δυνατότητες, γίνονται πιο οριζόντιες, λιγότερο αυθαίρετες οι δυνατότητες παροχής του εκπαιδευτικού υλικού του, του εκπαιδευτικού περιεχομένου και ξέρω ότι η κυρία Ροντρίγκες εδώ ετοιμάζει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το οποίο θα σας εντυπωσιάσει και καλύπτει τα θέματα αυτά. Πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια πιο ε, θετική ε, προσέγγιση, δυνατότητα υποδοχής και αποδοχής της γυναίκας ε, στο χώρο της εργασίας. Αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί. Πρέπει όμως να μιλήσουμε ιδιαίτερα για το θέμα της ε, συμμετοχής εκτός από την εκπαίδευση και στον επαγγελματικό βίο, τη δυνατότητα δηλαδή να στερεώνεται η παρουσία της γυναίκας στην κοινωνία όχι μόνο χάρη στη γνώση αλλά και στην συμμετοχή στο κοινωνικό γίγναστο και το επαγγελματικό. Έχουν λιγότερες ευκαιρίες όμως οι γυναίκες από τους άντρες και λιγότερες ευκαιρίες για επα, επικαιροποίηση των γνώσεών τους μέσω της διαρκούς κατάρτισης αντίθετα από τους άντρες. Αυτό λοιπόν η εδραίωση των γνώσεων έχει στρατηγικό χαρακτήρα, στρατηγική σημασία και εδώ θα σταματήσω και πρέπει να το συζητήσουμε παράλληλα με την οδηγία για την μητρότητα και την πατρότητα και επίσης υπάρχει ένα συμβολικό ε, μια συμβολική διάστηση ε, μέσα από τις προσπάθειες που γίνουν στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα θα υπάρξει άλλη μια ε, άλλο ένα μεγάλο άλμα που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και μιλάω για τη δική μου την πατρίδα, γιατί τη, γνωρίζω καλύτερα, αλλά δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Δηλαδή θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα ανυπόφορα εκείνα πρότυπα ανδρικής όσο και γυναικείας ταυτότητας, τα οποία αποτελούν, συνιστούν αμφισημεία, παραδείγματα και απώλεια προοπτικών, εσφαλμένες προσεγγίσεις δηλαδή, και αυτό θα πρέπει να το καταρρύψουμε. Το έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή των Γενικών άλλωστε. Και επίσης ε, στο συμβολικό πολιτιστικό επίπεδο πρέπει να δώσουμε περισσότερη θέση στις γυναίκες ε, με ένα πιο ανοιχτό ε, περιβάλλον επαγγελματικό. Σε αυτό πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρήσει. Πρέπει να εξασφαλιστεί δηλαδή ένα πεδίο, ένα περιβάλλον επαγγελματικό το οποίο να επιτρέπει το συγκερασμό του επαγγελματικού, του οικογενειακού βίου και όλων που αυτά συνεπιφέρουν. Όχι μόνο για του άντρε αλλά και για τι γυναίκε. Και ιδιαίτερα με το Women Economics που αποδεικνύει με τις μελέτες του ότι η απασχόληση των γυναικών έχει πολλαπλασιαστικό ρόλο για την εκπαίδευση των παιδιών, για την αύξηση του ΑΕΠ, και των πόρων, τη δημιουργία δηλαδή μια νέα ευημερία, αλλά επιπλέον δείχνει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν περισσότερο σε μικτές ομάδες, διοικητικά συμβούλια και το καθεξής, ή περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, στι γυναίκε, έχουν μεγαλύτερη επιτυχία χάρη στη δυνατότητά του να παράγουν καινοτομία. Αυτή είναι η νέα αποστολή που πρέπει να αναλάβουν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πολιτικές του νέου αιώνα. Αυτή είναι η δική μας, το, η δική σας η αποστολή. Ξέρουμε ότι μεγάλο κομμάτι του δρόμου έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως ακόμη. Και πάντως κάθε γενεά έχει το καθήκον να επανερμηνεύει και να προστατεύει τα όσα, να δεφυλάσει τα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχω πάθος για το θέμα αυτό. Σταματάω όμως για να δώσω το λόγο στους ειδικούς μας και τη συναλφοβουλευτή. Καταρχάς έχουμε την κυρία Στανίμιρα Χατζημίτοβα από την Βουλγαρία έχει ιδρύσει μια από τις πρώτες με κυβερνητικές οργανώσεις στην Βουλγαρία για τα θέματα της ότας των γυναικών, εκτελεστική διευθύντρια για πάνω από 40 project και συγχαρητήρια γι' αυτό στη χώρα της και την Νότια Ευρώπη. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και τους ε, ευρωβουλευτές και εθνικούς βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη σκέψη μου μετά από 20 χρόνια αφοσίωσης στον αγώνα της ισότητας των φίλων, ε, Αποφύτησα από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας και κατόπιν ε, πήρα πτυχίο οικονομίας. Και μετά την διάσκεψη του Πεκίνου άρχισα να ασχολούμαι με την ισότητα των ευκαιριών. Τότε μπήκε η ισότητα των δύο φύλων στη ψυχή μου και άλλαξε και τη ζωή μου. Η χειραφέτηση σημαίνει αξιοποίηση στο έπακρο του δυναμικού του καθενός. Και να αποφασίσουμε ότι η χειραφέτηση είναι ο πότερος σκοπός, η χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών είναι ο απότερο σκοπός μας και θα πρέπει να βάλουμε αυτή τη χειραφέτηση στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Επιπλέον θα πρέπει να επανεξετάσουμε, να επανεστιάσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη μόρφωση και την παιδεία. Είναι σημαντικό η αξιολόγηση να γίνει όχι μόνο στην πρωτοβάθμια, αλλά να συνεχιστεί και στη δευτεροβάθμια και την ανώτερη εκπαίδευση. Γιατί τι σημαίνει παιδεία, σημαίνει διαβίου εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση. Σημαίνει ε, συνειδητοποίηση, αφύπνιση και ευαισθητοποίηση στα θέματα της ισότητας των φύλων από το βρεφονιπιακό σταθμό, από την προσχολική ηλικία. Πριν από 10 χρόνια είχαμε ε, για 4 χρόνια ε, προγράμματα σπουδών με θέματα το, την ισότητα των φύλων σε σχολεία και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ήταν μια πολύ επιτυχής ε, δραστηριότητα το πρόγραμμα εκείνο. Βέβαια ε, αυτή η διαδικασία προϋποθέτει και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άρα κρατικές πολιτικές υπέρ της εμφυλίωσης της ε, οικογενειακής ζωής με τον επαγγελματικό βίο. Επανεστίαση, είπα προηγουμένως. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο ο αλφαβητισμός. Μας ενδιαφέρει η παγκόσμια ανάπτυξη, γιατί βρισκόμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Οπότε ε, η, η αγωγή του πολίτη, η δημιουργία αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμηση θα πρέπει να είναι τμήματα του προγράμματος σπουδών για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Για παράδειγμα, να αποτελέσουν αυτοπεποίθηση και για το σώμα τους τα κορίτσια. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δεξιότητες και των μαθητών και των, και των καθηγητών, ιδιαίτερα σε πολυεθνωτικές κοινότητες, να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα, το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν καλύτερα, να αναλύουν τις παγκόσμιες διαδικασίες, ε, να εξορθολογήσουν το ρόλο τους στο παγκόσμιο πλαίσιο για να γίνουν φορείς αλλαγής, ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου κόσμου. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε όλα αυτά, παρόλο που ο ορισμός της UNESCO για την παιδεία απαρτίζεται από τρεις πυλώνες, επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη. Ε, μερικές φορές η επίσημη εκπαίδευση επισκιάζει τις άλλες δραστηριότητες, οπότε η ανεπίσημη εκπαίδευση ε, μπορεί να συμβάλλει στην ε, υλοποίηση της ισότητας ε, και στην αηφορία της ισότητας, προκειμένου να ξεπεραστούν ε, οι διαφορές. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα σημεία. Στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, στην προσοχή που θα, θέσει, θα πρέπει να δώσουμε σε ιδιαίτερες ομάδες της κοινωνίας και στα δικά τους προβλήματα, Τρίτο θέμα, καθηγητές, δάσκαλοι, καθηγητές και τέταρτο, επενδύσεις, οικονομικές επενδύσεις στην παιδεία. Το σχολείο θα πρέπει να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Στο σχολείο θα πρέπει να καταρρύπτονται τα στερεότυπα των φύλων. Κάτι που δεν γίνεται, με ελάχιστες φαϊνές εξαιρέσεις στις σκανδιναβικές χώρες. Οπότε θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διαπαιδαγώγηση για τα δικαιώματα υγείας και σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών ε, και όχι κάποια μαθήματα θρησκευτικών που οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά εφόδια για να αντιμετωπίσουν τη σεξουαλική παρενόχληση μέσω του Ιντερνετ. 80% των θυμάτων είναι κορίτσια μεταξύ 11 και 16 ετών. Θα πρέπει να αναμίξουμε τα κορίτσια και τα αγόρια στην προσπάθεια της εξά, εξάλληψης της βίας λογοφύλου. Να μιλούμε φωναχτά για τη βία κατά των γυναικών. Θα πρέπει να δυναμώσουμε τις γυναίκες ε, για να αποτινάξουν το ρόλο του θύματος. Επίσης, να αποφύγουμε διακρίσεις ε, στην αγορά εργασίας, όπως ακούσαμε πολλές φορές σήμερα. Να δούμε τι έχουν μάθει οι γυναίκες, να δούμε ποιε είναι οι γνώσει τους και οι δεξιότητές τους για να τι προωθήσουμε στην αγορά εργασίας. Να εξασφαλίσουν έτσι μια οικονομική ανεξαρτησία και αργότερα, κάτι που δεν αναφέρθηκε ακόμη, να μπορέσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικούν και πολιτικά πόστα. Οι γυναίκε είναι φτωχότερε και δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τι προεκλογικέ του εκστρατείε το γνωρίζουμε και εσείς το γνωρίζετε θαυμάσια γιατί είστε πολιτικοί. Οπότε αυτή η αδυναμία των γυναικών ε, οδηγεί την, στην εξάρτησή τους ε, σε ηγέτες κομμάτων. Οπότε αναγκάζονται να υπακούν σε αυτούς. Για 9 χρόνια ε, συμμετείχα σε μια, συνεργάστηκα με συναδέλφου από την Task Force, την ειδική Task Force για την ε, πολιτική χειραφέτηση των γυναικών και είδαμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ακόμη και το σπουδάσουν οι γυναίκε, ε, δεν πληρώνονται ε, τόσο καλά όσο οι άνδρε και περιθωριοποιούνται στην αγορά εργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι νέε τεχνολογίε. Οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ποιότητα και ταυτόχρονα να προάγουμε την επιχειρηματικότητα ήδη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βλέπετε εδώ κάποια αριθμητικά στοιχεία. Δεν θα σταθώ σε αυτά γιατί πολλά ακούσαμε για αριθμητικά στοιχεία σήμερα. Αλλά θα σας μιλήσω για μία αναφορά που ξεκίνησε για την επευκαιρία της 8ης Μαρτίου από το Παγκόσμιο Ταμείο για τις Γυναίκες υπογρά... ε, προσυπέγραψα και εγώ αυτή την αίτηση που ε, προτείνει διάφορα μέτρα για να γεφυρωθεί αυτό το τεχνολογικό κενό μεταξύ των δύο φύλων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση των κοριτσιών και των γυναικών ε, στις επιστήμες ε, της τεχνολογίας. Και απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα επίπεδα εξουσίας ώστε να ξανάρθουν τα κορίτσια στο επίκεντρο της επιστήμης και της τεχνολογικής εξέλιξης. Θα πρέπει να έρθουν οι φραγμοί στην χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην μόρφωση και των κοριτσιών σε τέτοιου είδους τεχνολογικές σπουδές, αυξάνοντας την πρόσληψή τους και τη συμμετοχή του σε τέτοιε θετικέ επιστήμες και σε αντίστοιχε θέσει απασχόληση. Και επίση θα πρέπει και η επιστήμη και η τεχνολογία να ανταποκρίνεται στι ανάγκε των κοριτσιών και γυναικών. Αυτά προ τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Λίγα λόγια για την προσοχή που θα πρέπει να δώσουμε σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και στα δικά τους προβλήματα. Θα αναφερθώ κυρίως σε κάποιες εθνοτικές ομάδες και στους μετανάστες. Τι γίνεται με τους Ρωμά, τι γίνεται με τα κορίτσια και τις γυναίκες Ρωμά. Γνωρίζετε ότι είναι χαμηλότερο το επίπεδο μόρφωσής τους, ε, κατά πάσα πιθανότητα εγκαταλείπουν ε, και τη φίτηση, αφήνουν το σχολείο, έχουν άγνοια για τη σεξουαλικότητά τους, καμία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γι' αυτό και μένουν έγκες σε πολύ πρώιμη ηλικία, σε πολύ νεαρή ηλικία και επίσης έχουν και τα υψηλότερα ποσοστά αναλφαβητισμού τα κορίτσια Ρωμά. Κοιτάξτε τελευταία φράση της διαφάνειας. Ο διευθυντής του οργανισμού μας για την εθνοτική διαπαιδαγώγηση, διαπαιδαγώγηση εθνοτικών ομάδων, μου είπε ότι μεταξύ του 2004 και του 2014 παρατηρήθηκαν κάποιες θετικές αλλαγές στη Βουλγαρία. Οι γυναίκες Ρωμά έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ανώτατη εκπαίδευση και εγκαταλείπουν σε χαμηλ... λιγότερο το σχολείο. Και πάλι αναφέρθηκε από τη Διευθύντρια ότι 3.500 φοιτητές Ρωμά από 3.500 φοιτητές Ρωμά, οι 2.000 είναι φοιτητρίες, είναι γυναίκες Ρωμά. Πολύ σημαντική πρόοδος λοιπόν για τη Βουλγαρία. Λίγα λόγια για τους μετανάστες τώρα. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε ειδικά προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας ε, της χώρας υποδοχής και ίση πρόσβαση αγοριών και κοριτσιών σε αυτά τα μαθήματα. Επίσης ε, θέλουμε ε, ενθουσιώδεις καθηγητές, άνδρες και γυναίκες ε, καθηγητές και δασκάλους που θα είναι καταρτισμένοι σε θέματα ισότητας των δύο φύλων. Και θα πρέπει να εμπλέξουμε στον αγώνα αυτό και τους άνδρες, όχι μόνο τις γυναίκες. Και ξέρετε γιατί. Διαβάζοντας ε, το, τη σύνθεση της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντυπωσιάστηκα γιατί η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από, από 35 γυναίκες και δύο άντρες. Βέβαια το 50% των ανδρών είναι εδώ. Αλλά των ε, ανδρών ευρωβουλευτών της Επιτροπής ΦΑΜ δυστυχώς δεν είναι και το 50% των, ε, ευρω... των γυναικών ευρωβουλευτών της Επιτροπής ΦΑΜ. Επίσης, χρειαζόμαστε επενδύσεις στην μόρφωση, επενδύσεις στην παιδεία. Δυστυχώς δεν είναι καλές επιδόσεις της πατρίδας μου στα θέματα αυτά. 3,5% μόνο του ΑΕΠ δαπανίσαμε στην παιδεία μας, που είναι ανεπαρκέστατο ποσοστό. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι η ποιότητα είναι συνειφασμένη με την ε, οικουμενική πρόσβαση των ε, παιδιών σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Και επίσης ε, στο σχέδιο δράση, το για το 2015-2020 σε ό,τι αφορά την ισότητα των ευκαιριών, στην οποία συμμετέχει και η οργάνωσή μου, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί παιδεία που θα λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων και θα δίνει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν τις μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές αλλά και βέλτιστες πρακτικές με τρίτες χώρες. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Many, many thanks for this important... Και εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική σας εισήγηση και την έκθεση της εμπειρίας σας καθώς και για τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η δεύτερη, ο δεύτερος ηγητής για 10 λεπτά ή η κυρια Ζάλιγκερ που είναι ακτιβίστρια και εκπαιδεύτρια για την καταπολέμηση της βίας ε, κατά των γυναικών και έχει δημοσιεύσει διάφορα εγχειρίδια για την αυτοάμυνα των γυναικών. Uh, thank um, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για κάτι το οποίο εντάσσεται στο μη τυπικό κομμάτι της εκπαίδευσης Όπω είπε και η προηγούμενη μιλήτρια. Θέλω να σα μιλήσω για την φεμινιστική αυτοάμυνα. Θα ακούσετε τη λέξη φεμινιστικός πολύ από μένα, γιατί πιστεύω πως πρέπει όντω να επιτευχθεί η, η ισότητα των φύλων, αλλά χωρίς το φεμινισμό αυτό δεν γίνεται. Ε, αυτό σημαίνει ότι 110 χρόνια τώρα έχουμε ριζωμένες πεπιθήσεις μέσα στην ε, ε, παιδεία μας. Θέλουμε ωστόσο να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη των κοριτσιών απέναντι στην οικονομική πολιτιστική κατάσταση που μας κάνουν άνησες και που μας οδηγούν, οδηγούν μάλλον στην βία με βάση το φύλλο. Επίσης να αναζητήσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στις γυναίκες. Εφαρμόζουμε αρχές που προέρχονται από την φεμινιστική παιδαγωγική. Μία είναι η συνοχή ανάμεσα στους στόχους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Πράγμα που σημαίνει, εάν θες να εργαστείς για τη χειραφέτηση, θα πρέπει αυτό να το κάνεις επί εθελοντικής βάσης. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει τις γυναίκες και ε, τα κορίτσια να μάθουν πώς θα χειραφετηθούν. Αυτό έχει να κάνει με την αμφισβήτηση της ανισορροπίας των δυνάμεων εντός ε, ομάδων ανάμεσα σε καθηγητές και εκπαιδευτές. θα πρέπει να γνωρίζει κανείς και να είναι σε θέση να προβεί σε επιλογές ζωής και όλα αυτά σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ε, ζει. Έπειτα υπάρχει η μεροληπτική θέση ε, υπάρχει όμως ε, και το γεγονός ότι η γυναίκα θα πρέπει να είναι κύρια της ζωής της, υπεύθυνη και έτσι θα πρέπει να τοποθετηθούμε στο πλευρό των γυναικών και να τις βοηθήσουμε να υλοποιήσουν τις επιλογές τους. Ακόμα και αν εμείς προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούμε με αυτές τις επιλογές. το να είναι κανείς ε, φεμινιστής, ε, φεμινίστρια μάλλον ε, καθηγήτρια για την αυτοάμυνα σημαίνει ότι γενικά προωθώ την ισότητα των φύλων και πολύ σημαντικό τμήμα είναι η εκρίζωση κάθε συστήματος καταπίεσης όπως είναι ο ρατσισμός, η ταξική διάκριση, η ομοφοβία και όλες οι άλλες φοβίες που μπορεί να υπάρχουν ε, Δηλαδή είναι ο φεμινισμός ε, γενικός και ολοκληρωτικός. Εγώ είμαι ακτιβίστρια αλλά εργάζομαι σε μια πολύ μικρή οργάνωση εδώ στις, Γαλλί... στις Βρυξέλλες. Εργαζόμαστε με... Συνεργαζόμαστε με γαλλόφωνους, ολλανδόφωνους, αγγλόφωνους ε, ε, και η στόχος μας είναι η πρόληψη, η πρωτογενής πρόληψη της βίας με βάση το φύλλο, δηλαδή ό,τι μπορεί να κάνει κανείς πριν να συμβεί συμβεί η βία, πριν να υπάρξουν βία επεισόδια. Είμαστε μια μικρή ομάδα και αγωνιζόμαστε καθημερινά για να επιβιώσουμε, να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους μισθούς, να πάρουμε κάποια επιδότηση και να συμπληρώσουμε τις εκθέσεις και τις, τα έντυπα κτλ. Και είμαι βέβαια ότι στις περισσότερες χώρες που ε, αντιπροσωπεύετε εσείς εδώ υπάρχουν ένα σωρό τέτοιε ε, οργανώσεις που καθημερινά αγωνίζονται να επιβιώσουν, είναι, ανα, είναι αόρατες και δεν αναγνωρίζονται από κανέναν επίσημο θεσμό. Αυτό που κάνουμε είναι βέβαια μαθήματα αυτοάμυνας, αλλά όχι μόνο. Ε, δουλεύουμε για το θέμα του γενικού δημόσιου βήματος, ε, η αίσθηση ανασφάλειας. Προσπαθούμε να κάνουμε τις γυναίκες να αισθάνονται πιο ασφαλείς στην κοινωνία και να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χώρο, στο δημόσιο βήμα, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι ε, στο δρόμο. Και με όλα αυτά καταφέρνουμε να καταρτίζουμε πάνω από 700 γυναίκες και κορίτσια ετησίως και φτάνουμε σε πολύ περισσότερους από τους 700 που εκπαιδεύουμε διότι στα μαθήματά μας, εκτός από τα μαθήματά μας κάνουμε και δημοσιεύσεις αλλά και διασκέψεις και τέτοιου είδου ε, πράγματα. Τι, τι, είναι τώρα η φεμινιστική αυτοάμυνα. Όταν μιλάμε για αυτοάμυνα για τις γυναίκες, πολλοί σκέφτονται πολεμικές τέχνες. Δεν είναι ούτε καράτε, δεν είναι ούτε αϊκιντό, ούτε κλωτσοπατινάδα, ούτε τίποτα άλλο τέτοιο. Πάντως έχει να κάνει με το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, να έχει αυτοπεποίθηση και να έχει το δικαίωμα, να δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα να πει όχι και να κάνει τις δικές του επιλογές. Ένας ορισμός λοιπόν, γιατί υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, διάφορες μέθοδοι φεμινιστικής αυτοάμυνας, Πάντως ε, γενικά είναι οτιδήποτε κάνει τη ζωή ε, μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού πιο, ασφαλή και Περισσότεροι, οι ε, περισσότερα συστήματα περιλαμβάνουν τέσσερα βασικά συστατικά. Καταρχήν, κρίσιμη και σωστή ενημέρωση για τη βία κατά των γυναικών. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό μύθοι για το τι είναι η βία κατά των γυναικών, σε ποιον συμβαίνει, υπό ποιε συνθήκε, ποιοι είναι οι θήτε. Ε, και όλα ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν μας βοηθούν να προετοιμαστούμε και να προλάβουμε τη βία. Επίσης έχει να κάνει με στρατηγικές πρόληψεις, τι μπορεί να κάνει κανείς, τι λειτουργεί. Ε, πρέπει κανείς να γνωρίζει τα δικαιώματά του, τους νόμους που ισχύουν στην κοινωνία που ζει, τις υπηρεσίες που υπάρχουν ε, αν τις χρειαστείς. Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι οι τεχνικές ε, αυτοάμυνας. Ε, κάνουμε πολλές φορές ε, θέατρο και προσπαθούμε στην πράξη να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε σε καθημερινές καταστάσεις ε, όταν δεν γίνονται σεβαστά τα όρια μας ή όταν υποκείμεθα σε διακρίσεις, να, μπορούμε να πούμε τι δεν μας αρέσει και να, πώς να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να χτυπήσεις κάποιον θα χρειάζεται να συζητήσεις, να, να ξέρεις πώς να συζητήσεις για να σταματήσεις μια τέτοια κατάσταση. Φυσικά υπάρχει και, υπάρχουν και τεχνικές σωματικής άμυνας, απλές τεχνικές που είναι πολύ προσιτές. Μπορείς να τις μάθεις σε μια-δυο μέρες, αντίθετα από τις πολεμικές τέχνες. Δεν χρειάζεται χρόνια ε, προπόνησης για να μπορέσεις να τις χειριστείς. Αλλά πολύ σημαντική είναι και η ψυχολογική προετοιμασία που χρειάζεται κανείς για να ξεπεράσει τα εμπόδια τα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα στη διάρκεια της εκπαίδευσή μας ή της κοινωνικοποίησή μας για να σταματήσουμε να πούμε όχι εκεί που δεν θέλουμε κάτι και είναι απαραίτητο να πληγώσουμε κάποιον να είμαστε ε, ασφαλείς ωστόσο. Η φεμινιστική αυτοάμυνα δεν είναι προσωπική εξέλιξη ή ανάπτυξη, πρόκειται για συλλογική εκπαίδευση και αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών ανάμεσα στις γυναίκες, σε συλλογικών πρακτικών και επίσης είναι κομμάτι της αλληλεγγύης. Πολύ σημαντικό μήνυμα στα δικά μας μαθήματα είναι ότι αν θες να αλλάξει την κοινωνία στην οποία ζεις, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Θα πρέπει να προσπαθήσεις μαζί με άλλες γυναίκες για να καταφέρεις αυτές τις κοινωνικές αλλαγές. Αυτοάμυνα, η φεμινιστική αυτοάμυνα αφορά και την γνώση των ορίων του καθενός. Να είσαι σε θέση να πεις όχι και να δώσεις στον εαυτό σου το δικαίωμα να έχει όρια και να πει όχι. Τώρα, με τεχνικές σωματικής αυτοάμυνας, βλέπετε μία εδώ και έπειτα, επίσης θα πρέπει κανείς να σκεφτεί τι σημαίνει ασφάλεια, τι θα σήμαινε στις γυναίκες, για τις γυναίκες και τα κορίτσια και πώς μπορούν να το πετύχουν. Μεγάλο ερωτηματικό βέβαια είναι η πρόληψη αυτή λειτουργεί και τα καλά νέα είναι, ναι, λειτουργεί. Έχουν γίνει πολλές έρευνες από τη δεκαετία του 70 που δείχνουν Σαφώς ότι οι γυναίκες που αντιστέκονται στη βία πολύ συχνά καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που λειτουργεί καλά είναι το να αντιδράσει κανείς ε, νωρίς, να ακούσει την προέστησή του και να, μην, να αντιδράσει με δυσπιστία και θυμό και όχι με φόβο και δισταγμό και επίση πολύ σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιήσει κανείς μια μόνο στρατηγική, αλλά πολλές στρατηγικέ. Η πιο αποτελεσματική ε, στρατηγική είναι το να φωνάξει κανείς και να τρέξει να φύγει. Ε, εάν ένα μάθημα είναι ότι αν αντισταθείς, μάλλον οι γυναίκες σκέφτονται ότι αν αντισταθούν θα γίνει χειρότερα τα πράγματα. Όχι, η παθητικότητα είναι το μεγαλύτερο ρίσκο και αν αντισταθείς είτε προφορικά είτε σωματικά έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να ξεφύγεις με το λιγότερη ζημιά, μικρότερη ζημιά, η βλάβη. Επιπλέον όμως ε, της πρόληψης η φεμινιστική αυτοάμυνα έχει και άλλο αντίκτυπο. Υπάρχουν διάφορες έρευνες ε, που έχουν γίνει και που λένε, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν συμμετέχει σε τέτοια μαθήματα φεμινιστικής αυτοάμυνας έχουν καλύτερη ε, πάρκια ως προς τον εαυτό τους. Δηλαδή έχουν την πεποίθηση ότι μόνες τους μπορούν να χειριστούν τη ζωή τους, να αλλάξουν τη ζωή τους και να λάβουν αποφάσεις. Επίση, έχουν πιο συμμετοχικές διαδικασίε, είναι πιο ανεξάρτητες, ενώ ταυτόχρονα είναι λιγότερο φοβισμένε και έχουν λιγότερες από αυτέ τι συμπεριφορές αποφυγή που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία. Όπως για παράδειγμα το να μένουν σπίτια τους, να μην βγαίνουν εξωμόνες του ή να πηγαίνουν μόνο σε συγκεκριμένα μέρη γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι ασφαλή και ούτω καθεξής. Η αυτοάμυνα επίσης αυτού του τύπου επιβεβαιώνει και βελτιώνει την εικόνα που, έχει, που έχουν οι γυναίκες αυτές για τον εαυτό τους, την αυτοπεποίθησή τους, τις ε, δεξιότητες πρόληψης και χρησιμοποιείται και στην θεραπευτική ε, αγωγή μετά από την άσκηση βίας με βάση το φύλλο. Πολύ αποτελεσματική είναι λοιπόν η φεμινιστική αυτοάμυνα, αλλά χρειάζεται μεγάλη στήριξη και από την επίσημη πτυχή. Γιατί λοιπόν να μην μιλήσουμε για την αυτοάμυνα, για τα σχολεία, για τα κορίτσια μάλλον στα σχολεία. Στο επόμενο γύρο της συζήτησης περί εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να μην σωματωθεί η φεμινιστική αυτοάμυνα στις εθνικές δράσεις κατά της βίας κατά των γυναικών, η ε, των παιδιών. Επίσης είναι πολύ σημαντικό σε, να γίνεται σε χώρους μόνο για γυναίκες και πρέπει αυτούς τους χώρους να τους υπερασπιστούμε γιατί είναι χώροι ασφάλειας όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να συγκεντρωθούν, να σκεφτούν για την πραγματικότητα και να αναπτύξουν τις στρατηγικές που θα οδηγήσουν σε κοινωνικές αλλαγές. Και για να κλείσω την παρέμβασή μου θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτείτε πώς θα ήταν ο κόσμος αν κάθε κορίτσι και κάθε γυναίκα γνώριζε τον εαυτό της, τα όρια της και είχε δώσει στον εαυτό της το δικαίωμα να, έχει, να θέσει τα όρια της και να τα υπερασπιστεί. Αν κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι είχε τη δυνατότητα να πει όχι και να επιβάλλει το όχι της. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας ενδιαφέρουσες για μας. Και είναι και η άλλη όψη των ε, λεγόμενων υπείων ε, δεξιοτήτων που δεν είναι και τόσο ήπιες. Αναφερθήκατε στην διαχείριση των ε, συναισθημάτων και, συγκρούσεις, και συγκρούσεων. Πολύ σημαντικό ακόμη στοιχείο. Επίσης, τώρα προχωρώ για να δώσω το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο Λιλιάνα Ροντρίγκες για 10 λεπτά θα μας παρουσιάσει σε μερικές εβδομάδες μια έκθεση για τη χειρεφέτηση των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει βέβαια τον τελευταίο λόγο στη συζήτησή μας. Εγώ ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω για μια συνέντευξη τύπου με την Ιράτσι Τη δίνω το λόγο λοιπόν. Και τη διεύθυνση των εργασιών. Για να ολοκληρώσει. Έχουμε μόνο 15 λεπτά επιπλέον για τη διερμηνία και μετά θα πρέπει να κλείσετε. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Έχω μόνο 10 λεπτά στη θέση μου. Άρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κειμένου μου θα το αφήσω στην άκρη. Ήθελα όμως να σας παρουσιάσω τους στόχους μας και κάποιους πυλώνες από την έκθεση. Και θα μιλήσω πορτογαλικά. Είναι η μητρική μου γλώσσα και την προτιμώ. Ελπίζω ότι θα μας καλύψουν επαρκώς οι διερμηνείς. Ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη διοργάνωση, ευχαριστώ τους καλεσμένους του πάνελ. Θα κάνω μία νομική πλαισίωση, θα σας, παραφέρω, θα σας παραθέσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Η έκθεση που ανέλαβα θα μιλήσει για, την ισότητα των δύο φίλων και την προβολή της ισότητας αυτής, ε, τη χειραφέτηση, την ε, ανάληψη των ευθυνών ε, και την αντίληψη των δύο φίλων στην δημόσια και ιδιωτική ζωή. Η μόρφωση και η ίση πρόσβαση στην παιδεία θα πρέπει να ξεκινήσει όσο πιο νωρίς γίνεται στα σχολεία. Ακόμη και στο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή και στην προσχολική ηλικία. Και φυσικά θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συμπρόσβαση και αργότερα στη δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση. Η τελική μου έκθεση θα περιλαμβάνει τους εξής γενικούς στόχους. Πρώτος στόχος, η εξασφάλιση της ισότητας και της χειραφέτησης των κοριτσιών μέσω της παιδείας και της μόρφωσης. Δεύτερος στόχος, ελοποίηση της σύμβασης ε, της Κωνσταντινούπολης να ε, ε, ε, τα εκπαιδευτικά συστήματα με, κάποια, με κάποιους μηχανισμούς για τη χειραφέτηση και την αποφυγή της βίας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματική κουλτούρα ισότητας των δύο φύλων να ελέγξουμε τα προγράμματα σπουδών και τα, συνολικά, τα σχολικά βιβλία του να αναλαμβάνουν υπόψη, να λαμβάνουμε υπόψη τη ισότητα των ευκαιριών στη λήψη αποφάσεων προσωπικών και πολιτικών, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των γενικών σε ηγετικέ θέσει και στι θέσει και στις αγοράς εργασία και να προωθήσουμε την ισότητα και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να, να δούμε ποια είναι τα μέτρα που χρειάζονται για να υλοποιήσουμε αυτούς ε, τους στόχους που έθεσε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει να προωθήσουμε μπαθήματα ε, τεχνολογίας, επιστήμης, θετικών επιστημών και για τις γυναίκες, ε, να κάνουμε ενημερωτικές εκστρατείες για την άτυπη εκπαίδευση, να ελέγξουμε τα προγράμματα σπουδών και τα συνολικά βιβλία, να βελτιώσουμε την επιμόρφωση των καθηγητών υπό τη σκοπιά τη ισότητα των δύο φύλων και να κάνουμε μια γενική ευαισθητοποίηση και των γονέων στην ισότητα των δύο φύλων, προκειμένου να βελτιώσουμε την, και τη συμμετοχή των ανδρών στις ε, οικογενειακές ε, ευθύνες. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε και οικονομική στήριξη στις οικογένειες ε, για να προωθηθεί η αποστολή των κοριτσιών στα σχολεία για να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Θα προωθήσουμε λοιπόν τέτοιου είδους δράσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ θερμά τον Ευρωβουλευτή Μαραγκάλ για τη συμβολή του στην έκθεση είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε όλοι ώστε η παιδεία να λάβει υπόψη την ισότητα των δύο φύλων. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες της έκθεσης. Η κατάρτιση, το πρόγραμμα σποδών και τα σχολικά βιβλία. Τα μαθησιακά εγχειρίδια. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, ε, είναι σημαντικό να έχουμε νέες μορφές κατάρτισης ε, για την ισότητα. Θα πρέπει να έχουμε ε, αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση του δεκτικού προσωπικού, των ε, παιδιών, των νέων, των γονέων, των εργοδοτών, των εργαζομένων. Καλύτερη ενημέρωση λοιπόν της ισότητας των ευκαιριών και στις κοινότητες μέσω κοινοτικών οργανώσεων. Όπως είπε η Σίλβια, ε, δεν υπάρχει ουδέτερο σχολείο, όπως δεν υπάρχει και ουδέτερο πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών και να δώσουμε ανατολισμούς και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των δύο φύλων και η παιδαγωγική εποπτεία του προγράμματος σπουδών μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων. Ανάλυση και του άτυπου προγράμματος σπουδών. Εκεί θα πρέπει να προβλέψουμε επιπλέον δραστηριότητες που θα ενισχύουν το επίσημο πρόγραμμα σπουδών ε, ή ενισχύοντα την ισότητα των δύο φύλων. Δραστηριότητε που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών και τις εφοδιάζουν ε, με κάποιες ε, δεξιότητες όπως τα μαθήματα αυτοάμυνας αλλά και τεχνολογικές επιστημονικές γνώσεις ε, πλουτίζοντας τα εφόδια τους, τα πρακτικά και τα τεχνικά. Είναι σημαντική λοιπόν η κατάρτιση και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας για να ισχυθεί η επιχειρηματικότητα. Έχουμε και το άδειλο τώρα πρόγραμμα σπουδών σε αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, που δίνει έμφαση στις ε, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης. τέτοιου είδου άδειλο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να συνεργάζεται με τους καθηγητές ε, και σε επίπεδο αρχικής επιμόρφωσης και συνεχούς κατάρτισης. Εμπειρογνώμονες για την παιδεία και την ισότητα των φύλων θα πρέπει να προτείνονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αυτές, ε, αυτοί οι ερευνητές θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και να ενημερώνουν τους μαθητές και τους καθηγητές. Να αναλύουν δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών και να ενθαρρύνουν τους νέους για περισσότερη κοινωνική και πολιτική συμμετοχή. Θα πρέπει αυτή η κοινωνική συμμετοχή και η πολιτική συμμετοχή να ξεκινήσει ήδη από το σχολείο με την ενεργό συμμετοχή στα σχολικά συμβούλια, ενισχύοντας ε, την ε, ηγετική, τις ηγετικές ικανότητες των μαθητών. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση των κοριτσιών ε, στις θετικές επιστήμες και στις τεχνολογίες. Και να μην ξεχάσουμε και τις ποσοστώσεις ε, θα πρέπει να προβλέψουμε ποσοστό συμμετοχή των ανδρών στην ε, προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση που κυριαρχούνται κυρίως από γυναίκες. Επίσης, ε, για την κατάρτιση και την πληροφορία, γιατί μίλησα για τις κατά, για, τις, την αποφυγή του εκφοβισμού μέσω του ίντερνετ και οποιασδήποτε μορφής βίας ή παρενόχληση εντός και εκτός του σχολείου. Είναι σημαντική εταιρική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αρχών και μπορούμε με εσωτερικούς και εξωτερικούς ε, φορείς ε, να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε κατάλληλη εποπτεία και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών θα πρέπει να καταπολεμήσουμε στερεότυπα των δύο φύλων που θα... και μάλιστα α, ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία και συνεχίζοντας καθόλου τη διάρκεια της ζωής. Θα πρέπει να άρουμε τους φραγμούς στην πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας ή στην παρεμπόδιση των σωστών επιλογών. Επίσης, το δικαίωμα στη μητρότητα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει, το δικαίωμα στην πιτρότητα θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι εμπόδιο στην επαγγελματική σταδιοδρομία μιας γυναίκας. Αντίθετα θα πρέπει να θεωρηθεί ω ε, όφελος για ολόκληρη την κοινωνία. Και επίση θα πρέπει να προωθεί και, το, και η πατρότητα και η συμμετοχή και των ανδρών στι ε, οικογενειακέ υποχρεώσει. Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, επαναλαμβάνω, στα σχολικά βιβλία, στα, στα προγράμματα σπουδών και σε μεταγενέστερη αξιολόγηση από ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και εμπειρογνώμονε ισότητα ευκαιριών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολυκλαδικέ πολυκρατικέ ομάδε που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά βιβλία, εχειρίδια, ψηφιακό υλικό, επίση θα πρέπει να προωθεί την ισότητα των δύο φύλων και τη χρήση τη τεχνολογία από τα κορίτσια εντός του σχολείου. Επίσης, ε, να ε, ε, ελέγξουμε περιεχόμενο ανισότητα των δύο φύλων και εξάλληψη τέτοιου περιεχομένου από τα σχολικά βιβλία. Επίσης με το μαθησιακό υλικό θα πρέπει να προωθούμε την, την ισότητα ευκαιριών σε μικτές ομάδες που θα παρτίζονται και από μαθητές και από εκπαιδευτικούς. Έχουμε τέτοια εμπειρία στην Πορτογαλία. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τις δημοκρατικές αξίες και να θεωρήσουμε την ισότητα των φύλων ως κινητήριο μοχλό της κοινωνίας. Οπότε, σε καμία περίπτωση η, δική μου έκθεση, οποιαδήποτε άλλη έκθεση, ε, να μην ξεχνούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα των φύλων. Και γι' αυτό προτείνουμε να, να δημιουργηθεί και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ισότητας των Ευκαιριών στα Σχολεία. Και στείλουμε στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν τέτοιο βραβείο και εθνικά για να επιβραβεύεται το καλύτερο πρόγραμμα για την ισότητα των δύο φύλων. Γιατί μόνο με την ισότητα θα καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και την έλλειψη δημοκρατικότητας. Και σίγουρα τις επενδύσεις δεν είναι αντιφατικές με την πολιτική της ισότητας. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το επενδυτικό σχέδιο Juncker για τα κονδύλια αυτά, τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα, ευχαριστώντας τους άλλους, τις άλλες Με 10 μόνο, 15 λεπτά μόνο στη θέση μας. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι και όλες παρούσες. Ε, δύο λεπτά ο κάθε ομιλητής, κάθε ομιλήτρια. από την Ισπανία και το Κιντανίλε θα λάβει το λόγο μια μιλήτρια. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Ευρωβουλευτέ και Ευρωβουλευτέ, Θα ήθελα να συγχαρώ τους καλεσμένους ε, και τους εισηγητές και ειδικού ε, που έλαβαν μέρος σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα που εορτάζουμε την Διεθνή ημέρα της γυναίκας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλούμε λοιπόν για τη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών μέσω της μόρφωσης και της εκπαίδευσης. Ανοίξουμε μια ματιά στις χώρες μας, που είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνουμε ότι το 54% των γυναικών είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Στην Ισπανία το 60% των αποφύτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί να έχουμε τόσες πτυχιούχες δεν συμμετέχουν γυναίκες στη λήψη των αποφάσεων. Γιατί δεν συμμετέχουν πιο ενεργά στο εργατικό δυναμικό. Γιατί η μόνη τους πρωταγωνιστική θέση είναι στη γυναική ανεργία. Γιατί λείπουν ακόμη γυναίκες από τις ηγετικέ θέσεις. Πού αποτύχαμε στη διαπαιδαγώγηση της ισότητας και γιατί αυτές οι γυναίκες με πτυχίο πανεπιστημίου δεν μπορούν να φτάσουν στην αγορά εργασίας, στην οικονομία, στην πολιτική και δεν κρατούν τα ενία της ίδιας τους της ζωής. Σήμερα γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας. 40 χρόνια μετά την πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για τα δικαιώματα των γυναικών που έγινε στο Μεξικό. 20 χρόνια μετά την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη που έγινε στο Πεκίνο για τις γυναίκες. Πού αποτύχαμε και γιατί αποτύχαμε αποτύχαμε γιατί δεν εξασφαλίζουμε συμμετοχή των γυναικών ε, στη λήψη αποφάσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν σήμερα μια έκκληση προς, όλα τα, προς όλες τις κυβερνήσεις να χειραφετήσουν τις γυναίκες για να χειραφετηθεί η ανθρωπότητα. Περί αυτού πρόκειται. Όλοι μας, άνδρες και γυναίκες, που συμμετέχουμε σε επιτροπές δικαιωμάτων της γυναίκας και ισότητας των δύο φύλων στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συζητήσουν ε, το οριστικό κείμενο της πλατφόρμας του Πεκίνου και της, ε, ε, του θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει όλοι να υψώσουμε τη φωνή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιέχει το μήνυμα της Ένωσης την ξεκάθαρη δέσμευση της χειραφέτησης των γυναικών και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Γιατί το έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα σημαντικό κείμενο που όμως ε, δυστυχώς φέρει την υπογραφή οπισθοδρομικών χωρών που είναι κατά της πρόοδου των γυναικών. Γιατί υπάρχουν κυβερνήσεις απολύτως ανδροκρατούμενες κυβερνήσεις που δεν έχουν γυναίκες στα Υπουργεία τους θα ξεχάσουν τις γυναίκες και από τις πολιτικές τους. Ευχαριστώ. Και τώρα. Κυρία Κουτέλ, Γαλλία. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Μπερμπέρ. Η Γκέρμπερ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ θερμά για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Με, με εντυπωσιάζουν πάντα ε, διαπιστώσεις ότι πολλές φορές τα κορίτσια μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο μόνο και μόνο γιατί λείπουν ε, οι τουαλέτες, ε, οι εγκαταστάσεις υγιεινής. Αυτό βέβαια αφορά αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρώπη είναι δεδομένο την υποχρεωτική εκπαίδευση και έτσι εδώ έχουμε πιο πολύ να κοιτάξουμε προδιαγραφές και προσδοκίες. Τι περιμένουμε για τα παιδιά στο σχολείο έγινε λόγος για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση το πρωί. Είναι ζωτική σημασία για τα κορίτσια αλλά και για τα αγόρια. Γιατί αν τα αγόρια διδαχθούν ε, πώς ε, μπορούν να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους, ίσως να μην χρειάζεται ειδική ε, εκπαίδευση για τα κορίτσια σεξουαλική ή για την άμυνα, για την αυτοάμυνά τους. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ μεγάλη σημασία των ορμονών που σημαίνουν ορίμανση σε διαφορετικά στάδια, τα γόρια σε διαφορετικό στάδιο από, την, ε, από τα κορίτσια, οριμάζουν και μπορούν να μαθαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε σε χωριστά σχολεία. Δεν είναι αυτό η λύση. Πρέπει όμω να το χειριστούμε με έναν τρόπο πιο ευέλικτο μέσα στο εκπαιδευτικό μα σύστημα και να εξασφαλίσουμε μια κατάλληλη εκπαίδευση για τα κορίτσια και τα χώρια η συνεχιζόμενη, η διαρκή εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Εγώ σταμάτησα το σχολείο όταν ήμουν 15 ετών. Ο πατέρας μου θεώρησε ότι ήταν καλύτερο να με παντρέψει όταν ήμουν 15 ετών. Εγώ όμως τον διέψευσα. Λοιπόν, πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στα κορίτσια τα οποία χρειάστηκε προώρα να καταλήψουν το σχολείο με δουλειά και από τις οργανώσεις των ε, κοινοτήτων που είναι αυτές που υποφέρουν οι πρώτες από τις περικοπές βέβαια Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε αυτά ακριβώς τα πράγματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Και πρέπει να πω ότι εγώ τώρα που έχω εγκαταλείψει σχολείο μου στα 15 έχω γίνει ευρωβουλευτής. κυρία Μπέντζαμιν τώρα που είναι βουλευτής από την Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Εκπροσωπώ την Βούλη των Λόρδων, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης είμαι πρίτανης του Πανεπιστημίου του Έξιτερ ενός ε, πανεπιστημίου και μάλιστα μία από τις λιγότατες ε, πριτάνης πανεπιστημίων και η πρώτη μαύρη πρίτανης του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια και μίλησα για το χρώμα του δέρματος, βλέπω ότι υπάρχει μόνο άλλος ένας, άλλη μία ε, με προέλευση άλλη από τη Λευκή εδώ μέσα. Πρέπει αυτό να το σημειώσουμε και να προχωρήσουμε. Εμένα, η μητέρα μου όταν μεγάλωνα με τα άλλα τρία αγόρια και δύο κορίτσια, πέντε αδέλφια μου, ε, πάντα μας μάθαινε ότι πρέπει να δράξουμε τις ευκαιρίες μας στη ζωή. Αυτό μπορέσαμε να κάνουμε με την εκπαίδευση που μας άλλαξε τη ζωή, τη δική μας, αλλά μας επιτρέπει να αλλάξουμε και τη ζωή άλλων και μπορούμε χάρη στην εκπαίδευση να βελτιώσουμε τον τραυματισμένο αυτόν κόσμο. Αν μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, τότε μπορούν να φέρουν αυτή την αλλαγή που χρειάζεται στις, ε, και την ισορροπία στον κόσμο. Οι γυναίκες κάθε προέλευσης και υποβάθρου πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο τους για να προαγάγουν ένα κόσμο πιο ισορροπημένο, πιο δίκαιο έναν κόσμο στον οποίο όλοι θα αισθάνονται ότι έχουν τη θέση τους και την αξιοπρέπειά τους. Πρέπει και οι άντρες να αντιληφθούν ότι πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην προσπάθεια αυτή. Χρειάζεται η κατάρταση και ως προς σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις μεταξύ των φίλων για να σταματήσουν οι ανισότητες και η σεξουαλική βία. Ανησυχώ για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά ε, είναι εκτεθειμένα σε διαδικτυακή πορνογραφία εκεί που τη γυναίκα την παρουσιάζουν με έναν τρόπο εσφαλμένο και την μεταχειρίζονται με τρόπο εσφαλμένο. Η σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση νομίζω θα μπορέσει να φέρει μια αλλαγή νοοτροπία στα παιδιά μας. Θα τους διδάξει και η φιλοσοφία, η ανοχή, η αποδοχή, ο σεβασμός. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι πατάμε το κουμπί και αλλάζουμε σελίδα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που τηρήσατε και τα δύο λεπτά. Θα δώσω το λόγο τώρα στη Μέρη Μοράν από την Ιρλανδία. Thank Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να μιλήσω εδώ. Βρίσκω αυτή τη ε, διάσκεψη εξαιρετική και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τόσες γυναίκες παρούσες. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω έχουν ήδη υποθεί, αλλά δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε ακόμη περισσότερο τα ζητήματα τα οποία ήδη ε, τονίστηκαν σήμερα. Αν μπορούσα να μιλήσω για το Ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα που διορθωτικά τοποθετεί τα αγόρια και τα κορίτσια σε βάσει, βάσεις, ε, ωστόσο όπως και σε άλλες χώρες βλέπουμε το μίσο που τα κορίτσια υποαντιπροσωπεύονται και τα άλλους όπου τα αγόρια αντιστοίχως υποαντιπροσωπεύονται. Η σημερινή κυβέρνηση τονίζει μια πιο ουδέτερη ε, εκπαίδευση, ιδιαίτερα για τα παιδιά που δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Επάντω, εκεί που τα κορίτσια αντιπροσωπεύονται λιγότερο είναι οι θετικέ επιστήμες. Είναι ένα τομέας όπως και αλλού, όπου οι γυναίκε θα πρέπει να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στις, επιστημονικές, στις επιστήμες, στις τεχνολογίες, αλλά και στις, στη χαρτογράφηση. Εγώ έχω δουλέψει στην παιδεία Έχω μεγαλώσει και πέντε παιδιά ταυτόχρονα και μπήκα στην πολιτική πολύ πρόσφατα. Πρέπει πιστεύω να δώσουμε στις γυναίκες κάθε δυνατότητα, κάθε ευκαιρία να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ε, εκπαίδευσης. Ε, αν μου είχε πει κανεί πριν από τρία χρόνια ότι θα είχα την ευκαιρία να μιλήσω στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν, το είχα πιστέψει. Ε, αλλά αν δοθούν οι ευκαιρίες τι γυναίκες σίγουρα μπορούν να δράξουν την ευκαιρία και να σταθούν στο ύψο της περίσταση. Κάτι το οποίο έχει βελτιωθεί στην ισότητα των φύλων, τουλάχιστον στον απτυγμένο κόσμο, ε, είναι η ισότητα των φύλων. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι φραγμοί στην παιδεία για τις γυναίκες με παιδιά που θέλουν να επανέλθουν στην απασχόληση και όπως ε, υπόθηκε και προηγούμενα, η φροντίδα των παιδιών κοστίζει και είναι ένας μεγάλος φραγμός πέρα από το οικονομικό κόστος της επιστροφής στην εκπαίδευση. Ε, δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε επίσης το, ε, πόσο ωφέλιμο είναι για ε, τις πνευματικές της ικανότητες και την, και την αυτοπεποίθηση της γυναίκας. Η ισότητα των φύλων έχει μπει στην νομοθεσία μας στην Ιρλανδία. Αυτό ήταν σπουδαίο. Αυτή τη στιγμή 27 από 166 ε, βουλευτές γυναίκες και δεν νομίζω ότι η σχετική νομοθεσία θα βελτιώσει την κατάσταση. Και ζητώ συγγνώμη που λίγο ξεπέρασα το όριό μου. Θα σας δώσω τώρα όμως ένα λεπτό στον κάθε μιλητή γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Λιλιανά Μαρουσίκ, αν το είπα καλά, από τη Σερβία. Ευχαριστώ. Το σύστημα α, εκπαίδευσης της Σερβίας στηρίζεται στις, αρχές, στις εξής αρχές. Ισότητα πρόσβασης στην επιστήμη και στην ε, μόρφωση, πλήρως ε, σεβασμός των παιδιών, των ε, και των ε, παιδιών και των αγοριών και κοριτσιών και ίση ευκαιρία των ε, ίση ευκαιρία στην ε, κατάρτιση και στην παιδεία και των αναπήρων επίσης. Βασικός στόχος είναι η κατάργηση όλων των διακρίσεων και η υλοποίηση της ισότητας φύλων αλλά και της ισότητας μεταξύ των εθνοτήτων ισότητα και αποφύγει των διακρίσεων για λόγους φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και το καθεξής. Επίσης, έχουμε και νομοθεσία στα πλαίσια της προσπάθειας εκδημοκρατισμού που έγινε στη Σερβία και που τροποποίησε το εκπαιδευτικό σύστημα. Εκεί άλλαξαν βασικές διατάξεις, ε, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα των γυναικών και την ε, πρόσβασή τους ε, στην παιδεία. Έτσι προσπαθούμε να πραγματώσουμε μια κοινωνία της γνώσης που θα αξιοποιεί το δυναμικό και των ανδρών και των γυναικών. Έτσι θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της ε, Σερβίας ε, και της ε, κοινωνίας της Σερβίας αλλά και τη θέση της Σερβίας στον κόσμο με σεβασμό όλων αυτών των αρχών και των αξιών. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη κάλυψη του πληθυσμού σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία μέχρι την ανώτερη εκπαίδευση. Επίσης προβλέπουμε συνεχή και διαβίω κατάρτιση και εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς. Θέλουμε να εστενιστούμε τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Δυστυχώς πρέπει να κηρύξω το πέρας της συνεδρίασης, ευχαριστώντας σας θερμά για τη συμμετοχή και να σας καλέσω σε μια δεξίωση, σε ένα κοκτέιλ σεμνό στο δεύτερο όροφο του ίδιου κτηρίου. Γεια σας.